Καλημέρα σα, Θα μιλήσω ισπανικά. Σας δίνω λοιπόν λίγο χρόνο για να βάλετε τα ακουστικά σα. Μικρόφωνο παρακαλούμε για την Πρόεδρο. Καθώς ε, είναι κάπως φορτωσμένη η ημερήσια διάταξη και βιάζεται και είπατε εκπρόσωπο. Ε, θα ξεκινήσουμε γιατί έρχεται εκεί πρόεδρος, χωρίς χρονοτριβή λοιπόν. Θα αναλάβω εγώ την Προεδρία για λίγο και θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρούσο για να προβεί στην παρουσίασή του και το πρωτόκολλο και το καλωσορίζουμε θα το αφήσω στην κυρία Χολμάιερ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ρούσο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγητή και τα μέλη της Επιτροπής σας, ε, ε, αγαπητοί είπατε εκπρόσωπε τη εξωτερική πολιτική και της πολιτικής ασφάλειας. Χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα για να παρουσιάσω το κεφάλαιο 10 της ετήσιας έκθεσης του Ελεκτικού Συνεδρίου, την αξιολόγηση για τις διοικητικές δαπάνες, ιδιαίτερα σήμερα ε, σε ό,τι αφορά την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Το έτος 2018 οι πληρωμές δυνάμει του τομέα 5 του πολιτισμού δημοσιονομικού πλαισίου φτάνουν στα 9,9 δισεκατομμύρια ευρώ ή περίπου το 6,3% του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αξιολόγηση του ελεκτικού συνεδρίου στην ετήσια έκθεση 2018 είναι θετική και οι δαπάνες για τη διοίκηση δεν έχουν ουσιώδες φάλμα. Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται σε ένα δείγμα 45 συναλλαγών, από τις οποίες τέσσερις σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, δεν βρήκαμε καμία από τις συναλλαγές να διαπέτει από και επομένως δεν έχουμε συγκεκριμένες παρατηρήσεις ή συγκεκριμένες συστάσεις για την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Δεν ε, αξιολογήσαμε τη συνέχιση που δόθηκε στις γενικές μας συστάσεις που έγιναν προς την υπηρεσία στην ετήσια έκθεση του 2015, καθώς το ελεγκτικό μας έργο δεν κάλυψε τα είδη των συναλλαγών που σχετίζονται με αυτή. Πρόεδρε, ζητή, μέλη της Επιτροπής, παραμένω την διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις ή ερωτήσεις και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Καταρχήν ε, να σας ζητήσω συγγνώμη, γιατί ειλικρινά ε, μια ώρα χρειαζόταν για να έρθω εδώ. Ούτε καν το είχα φανταστεί ότι θα χρειαζόμουν τόσο πολύ χρόνο. Αλλά σε κάποιο σημείο έχουν ε, μπλοκάρει το δρόμο λόγω έργων και δυστυχώς δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Λυπάμαι πάρα πολύ που καθυστέρησα και ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφό μου που ξεκίνησε τη συνεδρίαση. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά την κυρία Μογκερίνη, την τη εκπρόσωπο. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα στη συνεδρίασή μας. Ε, η δική μας επιτροπή ε, ανέκαθεν σας εκτιμούσε ιδιαίτερα και θα ήθελα ευθύ αμέσω να σας δώσω το λόγο. Ε, δεν θέλω να σας καθυστερήσω γιατί ξέρω ότι μετά πρέπει να φύγετε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ τον κύριο Ρούσο. Δυστυχώς όπως όλοι φαντάζομαι πολύ καλά γνωρίζετε, πρέπει να πάω στην Ολομέλεια ε, για να τοποθετηθώ στα κατεπήγοντα σε περίπου 10 λεπτά, το πολύ 15 λεπτά. Ε, πρέπει να ε, δείξω ότι το σεβασμό μου για το Κοινοβούλιο, όχι μόνο για τις Επιτροπές αλλά και για την Ολομέλεια και ως εκ τούτου είμαι αναγκασμένη να αφήσω σε εσά τους συνεργάτες μου οι οποίοι θα απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις που ενδεχομένως έχετε. Αυτή είναι η έκτη διαδικασία απαλλαγής στην οποία συμμετέχω. Εγώ έχω θεωρήσει ανέκαθεν ότι η συνεργασία μας στον προπολογισμό για τις εξωτερικές δράσεις ήταν μια ευκαιρία ε, Όσοι από εσά ήσασταν κατά το παρελθόν στην Επιτροπή, θα γνωρίζετε ότι για μένα προφανώ ε, η απαλλαγή είναι ένα τεχνικό θέμα, αλλά είναι και μια ευκαιρία να συζητήσουμε με τα μέλη του Κοινοβουλίου πώ μπορούμε να βελτιώσουμε τι επενδύσει από τον προπολογισμό για εξωτερικέ δράσει. Και επίση αυτό που μα ενδιαφέρει είναι πώ ακριβώ ε, δουλεύουμε στην εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μικρό παράδειγμα. Όταν ξεκίνησα εγώ, οι ασκούμενοι δεν πληρώνονταν όσοι δούλευαν για την υπηρεσία εξωτερική δράση. Αυτό κατά την άποψή μου ήταν άδικο και ήταν και ε, αντικίνητρο για κάποιου που ήθελαν ενδεχομένω να έρθουν σε εμά. Έτσι λοιπόν θέλησα να διορθώσω αυτό το λάθος και επίση και την υπηρεσία μα να την καταστήσω όχι μόνο πιο δίκαιη αλλά και καλύτερης ποιότητας. Επίσης πρόγραμμα αμοιβόμενη εξάσκησης, ε, ένα εργαλείο για να έχουμε νέου δεσμού με του νέου ανθρώπου και με του τους μελλοντικούς ηγέτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Και 1,2 ε, εκατομμύρια ευρώ με τη βοήθεια του Κοινοβουλίου προβλέφτηκαν και εκταμιεύτηκαν για το 2018 και 1,6 εκατομμύρια για το 2019. Συνολικά 400 ε, ασκούμενοι οπεφελήθηκαν από το πρόγραμμα το 2018. Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξή σας ε, καθ' όλα αυτά τα αίτια από αυτήν την Επιτροπή. Το Κοινοβούλιο πάντα μας χορηγούσε την απαλλαγή στον προπολογισμό και θα ήθελα να ευχαριστώ και τον κύριο Πέτρο Ρούσο από το Ελεγκτικό Συνέδριο που είναι σήμερα κοντά μας και παρουσίασε αυτή την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2020 ε, και εκεί φαίνεται ότι το ποσοστό σφάλματος είναι πολύ χαμηλότερο ε, σε, για ε, αρκετά συναπτά έτη. Είμαι λοιπόν ε, πολύ ιδιαίτερα χαρούμενη για αυτό το επίτευγμα. Αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια είδαμε το ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο να αλλάζει. Άλλαξε πολύ περισσότερο από ό,τι μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε. Και ο προεπλογισμός κατά κάποιον τρόπο ακολουθεί αυτές τις αλλαγές που πρέπει να αντιμετωπίσουν και οι υπηρεσίες. αλλάζει ο ρόλος μας στον κόσμο και αλλάζει και η ανάγκη για περισσότερους πόρους. Σήμερα οι εταίροι μα ανά τον κόσμο περιμένουν από εμά να διαδραματίσουμε καθοδηγητικό ρόλο. Κατά κάποιον τρόπο είμαστε σημείο αναφορά ε, για πολλού ε, στον κόσμο. Παραδείγματο χάρη σε μια εποχή όπου βλέπουμε ότι ασκούνται όλο και περισσότερε πιέσει, εμεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήμασταν εκείνοι που μπορέσαμε να διασώσουμε το πολυμερέ σύστημα. Και αυτό δεν είναι μόνο δήλωση αρχών, αλλά είναι και η καθημερινή δουλειά που πρέπει να γίνεται. Πραγματικά σώσαμε τι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση από το να καταρρεύσουν. Εμεί βοηθήσαμε στο να εφαρμοστεί η πιο κρίσιμη πολυμερή συμφωνία όλων των εποχών, ε, συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, στόχοι της ε, χιλιετίας. Ε, αν ρωτήσετε κάποιον στην Αϊόρκη ή οποιονδήποτε άλλον ποιο ήταν πίσω από το να όχι μόνο να επιτευχθούν αυτέ οι συμφωνίε αλλά και να εφαρμόζονται, θα σα πούν αναμφισβήτητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα από την υποστήριξη προ τα Ηνωμένα ήμασταν και η ήρεμη φωνή σε περίοδου αντιπαράθεση. Στήριξαμε διαπραγματεύσει σε ολόκληρο τον κόσμο σταματήσαμε ε, πολλούς ε, πολιτείς πολέμους από την Κολομβία μέχρι τη Μοζαμβίκη και το πιο σημαντικό, εμείς στηρίξαμε την εφαρμογή γιατί γνωρίζουμε ότι μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και υπογραφή η Συμφωνία Ειρήνης, εκεί έρχονται τα πιο δύσκολα και ξέρουμε ότι αυτό είναι επένδυση και για τη δική μας την ασφάλεια γιατί ε, η επίλυση διαφορών τον κόσμο είναι σταθεροποιητικός παράγων για το εμπόριό μας, για τις κοινωνίες μας, για την ασφάλειά μας και ούτω καθεξής. Και κατόπιν ακολούθησαν εποχές όπου δεν υπήρχε περιθώριο για διάλογο και εκεί εργαστήκαμε για να προκύψει διάλογος. Παραδείγματος χάρη η ομάδα επαφών ε, με τη Βενεζουέλα. Έτσι λοιπόν καθ' όλα αυτά τα έτη οι εταίροι μας ε, μας εμπιστεύτηκαν, μπόρεσαν να βασιστούν σε εμά ως ε, ένα αξιόπιστο και συνεπή εταίρο. Ήμασταν σημείο αναφορά για εκείνους γιατί σε μια εποχή της παγκόσμιας σύγχυσης, να το πω έτσι πολύ ήπια, εμείς παραμείναμε πιστοί στις θεμελιώδεις αρχές μας. Και επίσης συστήσαμε και το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πακέτο, παραδείγματο χάνει για την Ουκρανία. Και σήμερα η χώρα αντίσταται περισσότερο βέβαια από ό,τι ήταν πριν από πέντε χρόνια. Αυτό όμω οφείλεται στη δική μα τη δουλειά. Και επίση ξεκινήσαμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων για την Αφρική. Επενδύουμε σε καλέ θέσει, βιώσιμε θέσει, κυρίω στι γυναίκε ε, στην Ήπειρο αυτή, έτσι ώστε η Ήπειρο και οι άνθρωποι τη να είναι πιο ισχυροί. Και αυτό ε, είναι πολύ είναι μεγάλο, ε, μα συμφέρει και εμά του Ευρωπαίου. Άρα, δηλαδή, το είναι παγκόσμιο σημείο αναφορά. Αυτό απαιτεί πολιτικέ ενότητα αλλά και και αυτά τα πέντε χρόνια νομίζω το Κοινοβούλιο το κατάλαβε αυτό πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη ημών αλλά και των προκατόχων στι πολιτικέ μα. ...σω λόγω του νέου ρόλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έχω προτείνει 30% αύξηση του προπολογισμού μα για τα επόμενα 7 έτη και χαίρομαι που η νέα Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει αυτή την πρόταση και ελπίζω να το στηρίξετε κι εσείς. Πέρα από του πόρου μα πρέπει να είμαστε και ε, μια πιο αποτελεσματική επαγγελματική υπηρεσία. Πιστεύω ότι τα πέντε χρόνια κατορθώσαμε να προσαρμόσουμε την υπηρεσία μα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Τέσσερα επιτέγματα θέλω να φέρω σύντομα καθ' όλα αυτά τα έτη. Θετικέ εξελίξει. Συνεργαστήκαμε ακολουθώντα τι προτάσει του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι αν τελικά προκύπτουν θετικέ εξελίξει στο να βελτιώνεται η ποιότητα και η μέθοδη εργασία ε, των υπηρεσιών μα, αυτό οφείλεται στην καλή συνεργασία τη δική μα υπηρεσία, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Κοινοβουλίου. Πρώτον, επεκτείναμε και εξυγχρονίσαμε το το δίκτυο των αντιπροσωπιών. Οι πρεσβείε μα εισαγωγικά, νομίζω κάπω έτσι μπορώ να τι πω, είναι ένα θεμελιώδη εργαλείο για την εξωτερική μα πολιτική, όχι μόνο γιατί μπορέσαμε να εργαστούμε για του Ευρωπαίου πολίτε σε πολλέ χώρε χώρες όπου πολλά κράτη-μέλη δεν έχουν διπλωματική εκπροσώπηση, δεν έχουμε του 28 σε όλα τα μέρη του κόσμου προφανώ, αλλά ε, εκπροσωπείται η Ένωση παντού, Το που σημαίνει ότι δεν βάζουμε μόνο μία σημαία, σημαντικό βέβαια και αυτό, αυτή την εποχή, αλλά είναι και ένας πολύ καλός τρόπος για να έχει κανείς καθημερινές επαφές με τις τοπικές αρχές, με τους τοπικούς συνομιλητές, όχι μόνο τους θεσμικούς αλλά και την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα, τα μέσα ενημέρωσης. Έτσι μπορούμε να εκπροσωπήσουμε τα συμφέροντά μας, να είμαστε γρήγοροι, πιο αποτελεσματικοί όταν προκύπτει κρίση ή να προλάβουμε κρίση. Το βλέπουμε αυτό επί τόπου. Όλα αυτά τα χρόνια άνοιξα τέσσερις νέες αντιπροσωπείες. Εφέτος μόνο ε, στο Τουρκμενιστάν και στο Κουβέιτ ε, και αυτές οι δύο χώρες είναι ένα τέλειο παράδειγμα ε, ε, το Τουρκμενιστάν στην Κεντρική Ασία, επεκτηνόμεθα εκεί, είναι καθοριστική σημασίας περιοχή, είναι η πύλη ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ανατολική Ασία και η νέα αυτή αντιπροσωπεία ε, κατέδειξε ότι είμαστε πολύ ισχυροί στην περιοχή, πολύ πιο ισχυροί από ό,τι θα ήθελαν οι εταίροι μας και εμείς επενδύουμε σε αυτό. Από την άλλη, όσον αφορά το Κουβέιτ στον κόλπο, είναι μια δύναμη ειρήνη, σοφίας και όπως ξέρετε εκεί υπάρχουν αυτή στιγμή πολλές εντάσεις, άρα μας συμφέρει να έχουμε ένα ανοιχτό διάλογο για τον, για ένα ανοιχτό διάβλο για διάλογο και συνεργασία σε καθημερινή βάση με την παρουσία επιτόπου. Το να επεκτείνουμε αυτό το δίκτυο των αντιπροσωπιών σημαίνει ότι η κοιτακτριά μας πρέπει να είναι ασφαλή για το προσωπικό μας. Επίσης πρέπει να σεμβόμαστε τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα και μετά ε, την ε, ε, σύσταση 2016 του ελεγκτικού συνεδρίου πλέον έχουμε ανοιχτό χώρο των με άλλα με άλλους εταίρους ε, και ε, καλύπτονται έτσι πλήρως οι δαπάνες. Κατόπιν τούτου νομίζω ότι τα 35 τετραγωνικά μέτρα ανά μέλος, ε, ανασυνεργάτια, αυτό το καλύπτουμε. Άρα δηλαδή οι συνεργάτες μας πρέπει να μπορούν να δουλεύουν με ασφάλεια. Οι περισσότεροι ζουν σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον και είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη που μας έχει προσφέρει το Κοινοβούλιο για να βελτιώσουμε την ασφάλεια στις αντιπροσωπείες. Παραδείγματος χάνει τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε περισσότερους ε, υπαλλήλου ασφαλείας, έχουμε ε, εξοπλισμένα οχήματα και επενδύουμε σε καλύτερα προστατευόμενα κτίρια. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επίση υποφελήθηκαν άμεσα από τον επαγγελματισμό των, των τοπικών ε, υπηρεσιών ασφαλεία με τι αποστολέ σα σε τρίτε χώρε. Άρα τα καταλαβαίνετε όλα αυτά πολύ καλά. Το δεύτερο που θέλω να πω αφορά σε υπαλλήλου που συνεργάζονται σε αντιπροσωπείς, κυρίω ε, στου τοπικού, ε, είναι δηλαδή οι μη υπήκοοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση που εργάζονται επί τόπου. Διαπιστώσαμε ότι οι κανόνε εργασία του είναι πάρα πολύ παλιοί, του 89. Όσοι δουλεύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν τα ίδια ατομικά δικαιώματα όπω οι συναδελφοί του που κάνουν ακριβώ την ίδια δουλειά, απλώ επειδή οι δικοί του εθνικοί ε, κανόνε είναι διαφορετικοί. Έτσι λοιπόν, εφέτο, με τη βοήθειά σα, αναθεωρήσαμε αυτό το θέμα και ε, προσφέρουμε καλύτερη κοινωνική ασφάλιση για του συναδέλφου μα. Ε, Παραδείγματο χάρη, έχουν ε, και δυνατότητα άδεια από 8 μέχρι 10 εβδομάδες. Άρα βλέπετε συνέπειες στις ευρωπαϊκές μας αξίες. Μιλάμε πάντα για τα δικαιώματα των εργαζομένων, για ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Ε, έχουμε πάνω από 3.000 επιτόπου εργαζόμενους ε, και Τώρα έχουμε τρει αποφάσει οι οποίε ελήφθησαν το καλοκαίρι, άρα δηλαδή σημαντική πρόοδο για τη ζωή τόσων πολλών ανθρώπων που υπηρετούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτο σημείο, η στρατηγική επικοινωνία. Αυτό είναι πολύ βαθιά στην καρδιά μου και στη δική σας με τη βοήθεια του Κοινοβουλίου. Τρεις task force για επικοινωνίες ε, για την ανατολική πλευρά, τα Δυτικά Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Ε, έχουμε λοιπόν περίπου 4.500 ε, περιπτώσεις ε, που εντοπίσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Η Υπηρεσία Στρατηγικής Πολιτικής έχει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, σημεία επαφή στα κράτη-μέλη, άρα δηλαδή είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίζουμε καλύτερα την προεκστρατεία της ενημέρωσης και με συντονισμένο τρόπο. Πέρα από την ενημέρωση, αυτές οι ομάδες κρούσης οργάνωσαν πολύ επιτυχημένες εκστρατείες ενημέρωση διοργανώσεις, παραδείγματος χάρη ε, για τη συνάντηση κορυφή ε, ανατολική ε, εταιρεία, για τη Συρία, για τα Δυτικά Βαλκάνια. Με αυτέ τι εκστρατείε, τα μηνύματά μα έφτασαν σε πραγματικά εκατομμύρια ανθρώπων στην Ευρώπη και εκτό αυτή. Και αυτό είναι το καλύτερο αντίδοτο στην, κακή, στην λάθος πληροφόρηση. Αυτό οφείλεται στην πολιτική αλλά και οικονομική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι σχετικά με το προσωπικό μα. Είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιό μα. Η ποιότητα, ε, τα κίνητρα, η αφοσίωση των συναδέλφων είναι εντυπωσιακή. Εγώ προσωπικά είχα την ευκαιρία να του αποχαιρετήσω στι αρχέ τη εβδομάδα και του είπα κάτι που θέλω να επαναλάβω και σε αυτή την επιτροπή. Ποτέ δεν είδα τόσο αφοσιωμένο προσωπικό, ε, ικανό, ε, διπλωματική υπηρεσία αλλά και η στρατιωτική υπάλληλοι, ποτέ δεν το είδα όσο εδώ σε αυτή την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι απαραίτητο για να διαδραματίζεται ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο. Και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να διασφαλίζουμε ότι θα κρατήσουμε τα καλύτερα ταλέντα από ολόκληρο τον κόσμο με ίσε ευκαιρίε για όλου. Η δουλειά που γίνεται για καλύτερη χρήση των εμπειρογνωμόνων από τα κράτη-μέλη και αυτό πρέπει να αναφερθεί. Έχουμε πάρα πολλού ε, που είναι αποσπασμένοι σε εμά, ε, κυρίω σε θέματα ασφάλεια και άμυνα και σε θέματα στρατηγική επικοινωνία. Επίση, μπορέσαμε κάποιους μη στρατιω... κάποιες μη στρατιωτικές θέσεις να τις μετατρέψουμε. Ε, αυτό όμως ε, που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι καταφέραμε να επιτύχουμε την ισορροπία των δύο φύλων στην υπηρεσία μας. Πολύ σημαντικό αυτό. Οι γυναίκες είναι περίπου οι μισές του προσωπικού μας. Εγώ όταν ανέλαβα ε, διαπίστωσα τότε ότι οι γυναίκες ήταν μόνο το 7% των ανώτατων θέσεων στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Σήμερα είμαι υπερήφανη ότι από τις 7 πήγαμε στο 27% το 27% των ανώτατων θέσεων είναι γυναίκες. Πριν από πέντε χρόνια ήταν το 22%. Σήμερα φτάσαμε ε, στη μέση, στους μεσαίους και στο 31%. Ε, έχουμε ακόμα πολλά. Όλα αυτά οφείλονται όμως στις ε, διαρθρωτικές αλλαγές που έλαβαν χώρα. Ε, χρησιμοποίησαμε δύο ομάδες κρούσης για τη σταδιοδρομία. Παρεπιπτόντως, επιτρέψτε μου να προσθέσω ως γυναίκα ε, ότι είναι δύσκολο το να μπορεί να συμβάσει κανείς την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. Δεν πρέπει να είμαστε βέβαια ικανοποιημένοι μέχρι να επιτύχουμε την πλήρη ισότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει έγιναν κάποια θεμελιώδη βήματα και τώρα έχουμε μια νέα γενιά γυναικών τόσο στις Βρυξέλλες αλλά και στις αντιπροσωπεία μας. Σε ηγετικές θέσει, ε, κυρίω σε μεσαίε θέσει, Αυτές οι γυναίκε είναι έτοιμες να αναλάβουν περισσότερε ευθύνε, και είμαι πεπισμένη ότι αυτή η δουλειά θα είναι καθοριστική ε, σημασία ε, για τι ίδιε και για να προχωρήσουν. Όλα αυτά τα χρόνια είδα με τα μάτια μου ε, την εξουσία και την, τη δύναμη και την ευθύνη που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα χέρια της. Ε, η πολιτική βούληση είναι καθοριστική για να μπορεί κανείς να εκμεταλλευτεί αυτό το δυναμικό ε, πλήρως και η πολιτική βούληση βεβαίως και αφορά αυτή την Επιτροπή. Πιστεύω λοιπόν ότι κυρίως σε αυτές τις εποχές και κλείνω με αυτό πρέπει να επιβεβαιώνουμε στους εταίρους μας αλλά και σε εμά τους Ευρωπαίους την θέλησή μας, την βούλησή μας να διαδραματίσουμε αυτό τον ρόλο που περιμένει ο κόσμος από εμάς. Το να είναι κανείς παγκόσμιος παίκτη για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Έχουμε τα εργαλεία, έχουμε τις ε, δυνατότητες, ε, υπάρχουν προσδοκίες και πιστεύω ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση, αν υπάρχουν πόροι, ε, είναι σημαντικό για μας και για τον υπόλοιπο κόσμο να είμαστε αποτελεσματικοί. Χαίρομαι που το καταλαβαίνει αυτό η νέα Επιτροπή, ο νέος ύπατος εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής ε, θα χειριστεί τα θέματα εξωτερικής πολιτικής ε, με επιτυχία. Είναι καλός μου φίλος ο κύριος Μπορέλ. Είμαι σίγουρη ότι η υπηρεσία είναι σε άριστα χέρια ε, και θέλω να πιστεύω ότι και εσείς θα συνεχίσετε να μας στηρίζετε όπως το κάνατε όλα αυτά τα χρόνια έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτυχθεί πλήρως, να παραμείνει παγκόσμιος παίκτη στον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Φοβάμαι ότι ήδη πρέπει να φύγω γιατί πρέπει να είμαι στην Ολομέλεια σε πέντε λεπτά. Ε, σας αφήνω στα, στους ικανούς μου συνεργάτες για να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας. Τελειώνω ευχαριστώντας όλους εσάς για τη δουλειά σας, για τη δουλειά που κάναμε μαζί. Καλή τύχη. Κυρία Μογκερίνη, εμείς είμαστε μια επιτροπή κυρίων και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για ό,τι κάνατε μέχρι τώρα και να σας ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στο μέλλον και στην Ολομέλη. And gentlewoman. Thank you for... Επιτροπή κυρίων και κυριών. Ωραία. Τώρα, ο Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι. Σίγουρα με ικανοποίηση θα ακούσατε τόσους θα ακούσετε τσεχικά, τόσα τσεχικά, δεν θα έχετε ακούσει ποτέ νομίζω σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Τέλος πάντων, είναι όμορφη γλώσσα τα τσεχικά οπότε εγώ στα τσεχικά θα σα εξηγήσω. Ήθελα βέβαια να χαρεί τα τσεχικά και η πατή εκπρόσωπο, αλλά εντάξει δεν είναι εδώ τι να κάνουμε. Θα σας μιλήσω λοιπόν για την απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Για αρκετό χρόνο μπορούσαμε να αλλάξουμε τα πράγματα, όχι και τόσο πολύ εν πάση περιπτώσει, πρόκειται για πέντε χρόνια για πέντε απαλλαγές από πλευρά τη Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμών. Θυμάμαι το 2016 για παράδειγμα, όπου θέλαμε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση να είναι πιο αποτελεσματική. Ε, οι ανώτεροι αξιωματούχοι να είναι πιο αποτελεσματικοί, να υπάρχει γεωγραφική ισορροπία, ισορροπία ε, μεταξύ των ε, φύλων, να υπάρξει μείωση 5% του προσωπικού, καλύτερη λογιστική διαχείριση. Το 2017 θέλαμε οι διοικητικές δαπάνες να χρησιμοποιηθούν καλύτερα. Θέλαμε επίσης απλοποίηση των γραμμών του προϋπολογισμού όσον αφορά τις δραστηριότητες της Ένωσης και γεωγραφική ισορροπία πάνω απ' όλα. Όπως επίσης βέβαια και ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων. Έτσι λοιπόν εξέτασα όλα αυτά τα αιτήματα που είχαμε τότε και νομίζω ότι τώρα ε, μπορούμε να πούμε ότι τα πήγε καλά η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Έχω όμως κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, ποιες είναι οι κύριες απειλές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το έργο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και έτσι να επηρεάσουν και τον αντίκτυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δρόμενα. Δεύτερον, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη γεωγραφική ισορροπία στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές όσον αφορά την εκπροσώπηση των χωρών μελών. Έχουμε 9 Βέλγους επικεφαλής αντιπροσωπιών, 15 ε, Γερμανούς, 16 Γάλλους και σε 21 θέσεις έχουμε Ιταλούς, ενώ έχουμε μόνο 5 Πολωνούς. Η Τσεχική Δημοκρατία, που είναι σε μέγεθος όπως και το Βέλγιο, έχει δύο επικεφαλής αντιπροσωπιών και η Ρουμανία έχει δύο, ενώ είναι πολύ μεγαλύτερη. Το Βέλγιο έχει 18, η Γαλλία 35, και άλλες χώρες πολύ λιγότερους. Έχουμε δεδομένα επίση για τις δαπάνε όσον αφορά τα κτίρια. Πάντω για μένα και τους κοιόδης εισηγητέ είναι ασαφές που ακριβώς πάνε οι δαπάνε αυτές. Από ό,τι κατάλαβα, ε, κάποιες ε, μισθώσεις για κτίρια έχουν κοστίσει ε, πάρα πολλά χρήματα στο Λίβανο, στην Ταϊλάνδη, όπως επίσης και διαμερίσματα στην Κολομβία, την Αίγυπτο και το Χονγκ κάποιοι από τους λογαριασμούς που μας έχουν έρθει είναι πάρα πολύ ψηλοί, οπότε θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι υπάρχει πίσω από τις δαπάνες αυτές. Έπειτα για να μπορέσουμε ε, να περάσουμε στην επόμενη απαλλαγή, θα θέλαμε να ξέρουμε και το πλαίσιο των δαπανών αυτών. Νομίζω ότι αυτό θα βοηθούσε να έχουμε ακόμα καλύτερο διάλογο από αυτόν που ήδη έχουμε. Έπειτα το θέμα της ασφάλειας των κτηρίων και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Θέλουμε να ξέρουμε τι σχέδια έχετε για το μέλλον στον τομέα ακριβώς της ε, ασφάλειας και προστασίας. Και τέλος, και αυτή είναι μια προσωπική δική μου ερώτηση, για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και τις δομές διαχείρισης που έχει. Εσείς Πώς εκτιμάτε τη συνεργασία σας με τη δικιά μας Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μου επιτρέψετε να δώσω ευθύς αμέσως το λόγο στο Γενικό Διευθυντή. Ε, okay, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Θα ξεκινήσω από το τέλος, από την τελευταία σας ερώτηση όσον αφορά τη συνεργασία που έχουμε με την Επιτροπή σας. Ήταν καλή, πάρα πολύ καλή θα έλεγα όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι θέμα όχι τόσο δομή όσο θέμα ανδρών και γυναικών που συνεργάζονται. Για μας είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε ε, να σκεφτούμε διαφορετικά, να ακούσουμε πράγματα τα οποία ίσω εμεί δεν σκεφτόμαστε, επειδή εμεί είμαστε στι διαδικασίε αυτέ σε καθημερινή βάση. Οπότε είμαι πραγματικά ευγνώμων για την συνεργασία ε, που είχαμε μέχρι τώρα μαζί και που είμαι σίγουρο θα έχουμε και στο μέλλον. Τώρα έρχομαι στι επιμέρου ερωτήσει σα. Πρώτον, για τη γεωγραφική ισορροπία. Ναι, προσπαθούμε να πετύχουμε καλύτερη ισορροπία με την εκπροσώπηση και των νέων χωρών μελών, όχι μόνο ε, των παλαιών, ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Το 2018, 21% ήταν οι παλιές χώρες και 79, ε, ήταν οι καινούριες χώρες και το 79% ήταν από τις παλιές χώρες. Κάτι το οποίο ευθυγραμμίζεται κάπως ε, με την αντιστοιχία του πληθυσμού των χωρών των παλαιών και των νέων. Και αυτό για όλες τις κατηγορίες με κάποιες εξαιρέσεις στην Κύπρο. Από την Κύπρο για παράδειγμα δεν είχαμε ε, διπλωματικό. Κάτι το οποίο άλλαξε το 2019 γιατί ούτε από τους Δανούς δεν είχαμε τώρα. Έχουμε και Κύπριους έχουμε διπλωμάτες που εντάσσονται ε, στην υπηρεσία μας. Όσον αφορά τώρα τις ε, θέσεις ε, επικεφαλής αντιπροσωπιών πετύχαμε να έχουμε δύο από την Κύπρο που δεν είχαμε πριν και ελπίζουμε να έχουμε και Κροάτες την επόμενη φορά που δεν είχαμε μέχρι τώρα. Πρέπει επίσης να δούμε πώς δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, η οποία δημιουργήθηκε το 2010 με απόφαση του Συμβουλίου. Με προσωπικό από τις ήδη υπάρχουσες δομές, από την Relax, Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο που προσελκύσαμε τότε. Έτυχε να είναι πολύ Ιταλοί, τότε Γάλλοι, Βέλγοι κλπ. Οι συνάδελφοι αυτοί ε, παραμένουν, έχουν ε, μια σταδιοδρομία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Επίσης, τότε είχαμε και 120 νέες θέσεις. Δυστυχώς όμως, εξαιτία της κατανομής που ανέφερε και ο εισηγητής, έπρεπε να επιστρέψουμε 84, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα περιθώρια ελιγμών που είχαμε. Τώρα, οι προσλήψει είναι βάση αξιοκρατίας για τις υψηλές θέσεις επικεφαλής αντιπροσωπιών, για παράδειγμα, ή άλλες. έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία προσλήψεων με δημοσίευση που γίνεται εκτός και εντός του οργάνου. Έχουμε μια σύνθεση που απορρέει από το Γενικό Συμβούλιο, από, το, από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ε, και της Επιτροπής για να επιλέγονται οι υποψήφοι. φτάνουμε στην ύπατη εκπρόσωπο, η οποία παίρνει και την τελική απόφαση. Πάντως γίνεται πάρα πολύ σοβαρά αυτή η δουλειά. Τώρα για να προωθήσουμε τη γεωγραφική ισορροπία δύο πράγματα. Πρώτον, ο πληθυσμός γυράσκει. Εννοείται ότι οι υπάλληλοι από τις πρώτες 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεγαλώνουν, γερνάνε. Έχουμε ένα δίκτυο διευθυντών που συναντιέται τρεις φορές το χρόνο και προτείνει, μάλλον ζητάει να προτείνουμε ε, υποψηφίους για να καλυφθούν ε, οι θέσεις. Μερικές φορές για 43 ε, θέσεις έχεις πολύ λίγους. Προσπαθούμε λοιπόν να είμαστε σε επαφή με τα Υπουργεία στις χώρες μέλη και να τους προσελκύσουμε με διάφορες πολιτικές. Να, όπως είπε και η ύπατη εκπρόσωπος, να βοηθάμε να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή, για να έχουμε και ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων. Αυτά τώρα για τις διαφορές όσον αφορά την ισορροπία. Τώρα όσον αφορά την κτηριακή πολιτική που είναι και αυτό κάτι πολύ σημαντικό και το γνωρίζει η Πρόεδρος ε, καλά. Κάναμε πολλές προσπάθειες. Τώρα είμαστε στην διαδικασία όπου αναλύουμε με το ελεγκτικό συνέδριο ε, την έκθεση για την κτηριακή μας πολιτική. Νομίζω ότι είχαμε απόλυτη διαφάνεια, δώσαμε όλα τα στοιχεία που μας ζητήσατε. Ε, φυσικά χρειάζονται ερμηνεία αυτά τα στοιχεία. Πάντως να ξέρετε ότι απόφαση για τα κτίρια βασίζεται σε διάφορους παράγοντες. Τη σταθερότητα, τι αγοράζουμε, τι νοικιάζουμε, ανάλογα με την κατάσταση, ανάλογα με τη χώρα, αν θα μείνουμε για πάντα ή όχι, αν ε, βρίσκουμε καλές ευκαιρίες στην αγορά ή όχι. Η προβολή, γιατί θέλουμε εννοείται να προβάλλουμε την ε, διπλωματική ε, αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν μοιραζόμαστε το κτίριο με την ΕΚΟ ή με κάποιο άλλο οργανισμό. Και το πιο σημαντικό βέβαια είναι η ασφάλεια και η προστασία του προσωπικού μας. Συνεπώς δεν είναι εύκολο να εξηγήσει κανείς έτσι τώρα την κατάσταση. Φυσικά με λεπτομέρειες άμα θέλετε να συναντηθούμε μεταξύ μας και να σας δώσουμε όλες τις λεπτομέρειες. Τώρα για το Λίβανο. Φυσικά και είναι μια σημαντική αντιπροσωπή και έχουμε 87 ε, προσωπικό. Έχουμε το κτίριο μαζί με την ΕΚΟ εκεί. Και 3.290 τετραγωνικά μέτρα είναι το κτίριο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πληρώνουμε 330 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, κάτι το οποίο είναι κάτω από το μέσο όρο αλλά είναι και κτίριο με ασφάλεια. Εννοείται ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε την κάθε περίπτωση χωριστά και δεν έχουμε τώρα ούτε το χρόνο ούτε την ευκαιρία να το κάνουμε. Αλλά σημειώνω την ερώτησή σας ότι θέλετε περισσότερες πληροφορίες. Τώρα, για την ασφάλεια. Είναι κάτι το οποίο προσέχει πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε επιτελέσει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν ε, οι υπηρεσίε μα στο Δουβλίνο, για παράδειγμα, ε, που ασχολούνται με το θέμα αυτό, ε, δίνουν κατάρτιση στους επικεφαλείς των αντιπροσωπιών, ώστε να υιοθετούν τα κατάλληλα μέτρα. και τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Έχουμε και τη στήριξη των δημοσιονομικών αρχών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήθελε πάρα πολύ να το πετύχουμε. Πάντως το θέμα της ασφάλειας δεν είναι μόνο η δυνατότητα που έχουμε να δράσουμε επί τόπου, είναι και θα έλεγα η προστασία όλων Γίνεται λοιπόν μεγάλη προσπάθεια κατάρτισης του κόσμου που βρίσκεται στις διάφορες αντιπροσωπείες μας και το 99% του προσωπικού περνάει από κατάρτιση πριν πάει σε αντιπροσωπείες. Έχουμε επίσης και εκστρατείες συνειδητοποίησης επιτόπου. Όλες οι αντιπροσωπείες έχουν ένα τέλεχος που ασχολείται με το θέμα αυτό. Έχουμε κανόνες ε, για κένωση κτίριων κλπ. κλπ. Το θέμα της ασφάλειας πρέπει να το δούμε πέρα από την φυσική προστασία των ατόμων. Έχει να κάνει και με τις πληροφορίες και με την ασφάλεια των δικών μας ανακοινώσεων. Ξέρετε, το στοιχείο κλειδί είναι ότι προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια των δικτύων μας. Και προς το παρόν έχουμε καλύψει το 60% του δικτύου, προχωράμε όμως περισσότερο και το 2020. Με σύστημα ε, για εμπιστευτικές πληροφορίες. Συνεργαζόμαστε επίσης σε χαμηλότερο επίπεδο για ε, πιστευτικές πληροφορίες και ανακοινώσεις και με διάφορες εφαρμογές ε, στο κινητό ώστε να προστατεύονται οι πιστευτικές μας πληροφορίες. Και εδώ συνδυαζόμαστε και με το Συμβούλιο και με την Επιτροπή ώστε το μελλοντικό μας δίκτυο ασφάλειας επικοινωνίας να συνδυαστεί μαζί τους. Επίσης, δεν αφορά μόνο τις χώρες μέλη, αφορά και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης η ασφάλεια αυτή. Πρέπει να είμαστε ειδικοί εμπειρογνώμονες σε θέματα επικοινωνιών, σε θέματα πληροφοριών, σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Εννοείται ότι δεν κάνουμε ανοιχτό διαγωνισμό. Το 2021 θα επανέλθουμε και σίγουρα θα έχουμε βελτιώσει την προστασία, εφόσον βέβαια έχουμε τους κατάλληλους πόρους για να προσλάβουμε και τους κατάλληλους εμπειρογνώμονες. Είναι κάτι που αφορά όλες τις χώρες μέλη. Και θα έλεγα ότι είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος το θέμα αυτό της ε, πληροφορίας, που, στο οποίο αναφέρθηκε και είπατε εκπρόσωπος εξάλλου. Σας ευχαριστώ θερμά ε, για την ε, διεξοδική απάντησή σας και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους ε, σκιώδεις εισηγητές, αλλά να έχει την καλοσύνη να μην ξεπεράσετε τα πέντε λεπτά, γιατί αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα χρόνου. Η πρώτη είναι η Ιζαμπέλ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να μην μιλήσω καν πέντε λεπτά. Θα ήθελα να ξεκινήσω σχολιάζοντας το πόσο λεπτομερείς απαντήσεις δώσατε στο αριθμητολόγιο της Επιτροπής αυτής. Όμως, μου ανέκυψε μια σειρά ερωτήσεων βάσει των απαντήσεων που δώσατε. Καταρχήν, θα ήθελα να μου πείτε αν ε, η δημοσκόπηση του προσωπικού το 2018 μας έδωσε σημαντικά αποτελέσματα που θα μπορούσαν να συσχετιστούν με ε, τις περικοπές του 5% στο προσωπικό του 2014 και αναφέρουμε σε θέματα burnout, stress ε, ή υλοποίηση καθηκόντων που αντιστοιχούν σε ανώτερους. Η κυρία Μογκερίνη ανέφερε την ε, αύξηση σε ενδιάμεσες και σε υψηλές θέσεις. Όμως ε, θα ήθελα να μου πείτε ποιες ε, άλλες δράσεις πέρα από τη συγκεκριμένη κατάρτιση υλοποιεί υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, για να αυξήσει τον αριθμό των γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις και επίσης τι σημαίνει στο εσωτερικό της υπηρεσίας σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα πρακτικών στις ε, αντιπροσωπείες. Αν μπορείτε να μας πείτε ότι αυτοί που λαμβάνουν υποτροφίες ε, και οι που είναι υποχρεωτική πρακτική, αν λαμβάνουν ε, κάποια στήριξη, κάποια βοήθεια από την πλευρά της υπηρεσίας και αν υπάρχει κάποια εξήγηση υπορριθμών των υποτρόφων των έχει φτάσει από 26 σε 109 το 2018 σε ό,τι αφορά το δίκτυο συμβουλών ε, του έμπιστου προσωπικού. Ποια συγκεκριμένη κατάρτιση λαμβάνουν οι σύμβουλοι αυτοί, αν ε, δέχονται και ψυχολογική υποστήριξη και πώς η υπηρεσία διασφαλίζει ότι σέβονται το απόρριτο των δεδομένων, το χάρη όταν ανταλλάσσουν ε, στο δίκτυο πληροφορίε ε, και γιατί έχουμε μόνο τόσου συμβούλου από τι 140 αντιπροσωπείε ε, και διευκρινίζεται ότι μπορούν να ασχολούνται με θέματα που φορούν άλλε αντιπροσωπείε για να μην υπάρχουν συγκρούσει συμφερόντων. Δεν πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει προδραστική εστίαση από του συμβούλου σε σχέση με του συναδέλφου του αν θέλουν να αποφύγουν τη σύγκρουση συμφερόντων ενώ ταυτόχρονα ταυτόχρονα ε, διατηρείται ο παράγοντας της εγκύτητας μεταξύ των συμβούλων. Ich darf den nächsten Schattenberichterstatter bitten. Επόμενος και ο συγητής, ε, συνάδελφος Κινέα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θα αναφερθώ στο θέμα των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη δέχονται επίθεση σε τέτοιο επίπεδο. Υπάρχει ε, ένας ε, μηχανισμός προπαγάνδας από τη Ρωσία και από ΜΜΕ ε, που χρηματοδοτούνται από το κράτος και οι χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης είναι ακόμη πιο ευάλωτες σε τέτοιες επιθέσεις. Και βλέπω αυτό το πρόβλημα και το πώς απαντούμε. Παραδείγματο χάρη, βλέπω στις γραπτές σας απαντήσεις ε, ότι το East Stratcom Task ε, είχε αυξημένο προπολογισμό από 1 εκατομμύριο σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Όμω αυτό είναι γελίο σε σχέση με την σοβαρότητα του προβλήματος. Το σχέδιο δράσης ήταν ένα καλό βήμα προς τα μπρο, όμως η ερώτησή μου είναι περισσότερο πολιτικής και ελπίζουμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα για το μέλλον. Πιστεύετε ότι ω Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε του κατάλληλου όρου, επενδύουμε αρκετά για να καταπολεμήσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα και τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο κ. Κινέα και έρχεται συνάδελφο Πέξα, αλλά δεν θέλει να λάβει το λόγο. Ο κύριος Κούς. Ε, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Χολμάια. Εγώ έχω κάποιες ε, ερωτήσεις ε, γενικής φύσεως. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο το γεγονός ότι το ελεγκτικό συνέδριο δεν βρίσκει ουσιώδη σφάλματα. Όταν πρόκειται για έναν τέτοιο οργανισμό, μιλάμε για περίπου 10 δις ευρώ που εκταμιεύονται, είναι βέβαια αυτό εντυπωσιακό πρέπει να πω. Εγώ δούλεψα πάρα πολλά χρόνια στον ε, έλεγχο των οικονομικών. Ε, κατά κανόνα πάντα κάτι βρίσκουμε. Γι' αυτό λοιπόν διαρωτώ αυτό το ουσιώδες φάλμα. πώς ακριβώς ορίζεται και μήπως υπάρχουν τουλάχιστον τυπικά λάθη. Αυτή κυρίως είναι μια ερώτηση που στο ελεγκτικό συνέδριο όπου παραδείγματο χάρη είναι στα επαγγελματικά ταξίδια. Υπάρχουν χιλιάδε επαγγελματικά ταξίδια. Εκεί δεν μπορεί να μην υπάρχουν κάποια λάθη. Ή ε, στην αγορά των αυτοκινήτων. Και εκεί κάποια λάθη θα έχουν παρισφρήσει. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Και το άλλο μου ερώτημα αφορά στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Εσείς ε, Πώς τα καταφέρνετε έτσι ώστε να μην εμφανίζονται ουσιώδη σφάλματα. Ε, πώς το καταφέρετε αυτό. Ε, έχετε δικό σας ε, εσωτερικό έλεγχο ή παραδείγματο χάρη σε όλες αυτές τις αλλαγές προσωπικού που αναφέρθηκαν. Εκεί στις αλλαγές προσωπικού δεν κάνετε ε, καταγγελίες συμβάσεων. Δεν ακολουθούν διαδικασίες μετά από αυτές τις καταγγελίες και αν ναι, γιατί η υπηρεσία εξωτερικής δράσης τελικά, αν δουλεύει με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να μην εμφανίζεται κανένα, μα απολύτω κανένα ουσιώδε φάλμα, τότε αυτό θα πρέπει να είναι benchmark για όλου του άλλου θεσμού. Ε, σημείο αναφορά και σύγκριση. Θα ήταν δηλαδή καταπληκτικό. Αλλά ξέρετε κάτι, επειδή έχετε τόσε πολλέ δραστηριότητε και αλλαγέ, δεν ξέρω, εγώ δεν το πολύ πιστεύω αυτό που μα είπατε, πρόεδρο. Ε, συνάδελφε Κού, ε, να σα πω ευθύ εξ αρχή ότι η υπηρεσία εξωτερική δράση είναι κάτω από το κατόφλι εκείνου που το αντιμετωπίζουμε με κριτικό τρόπο. Είναι δηλαδή κάτω από το 2%. Τώρα, στο το ότι στην υπηρεσία εξωτερική δράση ε, δεν υπάρχει κανένα, μα απολύτω κανένα σφάλμα, δηλαδή 0,00. Ε, εντάξει, δεν το είπε κανεί αυτό. Ναι, αλλά το γράψατε όμω. Σας λέω, λέει η Πρόεδρος, επαναλαμβάνω, είναι κάτω από το 2%. Το 2% ορίζουμε ως κατόφλι ουσιώδου σφάλματος. Άρα γι' αυτό μάλλον κάπως ε, δεν το ορίσαμε σωστά. Προφανώς υπάρχουν κάποια σφάλματα. Από τη στιγμή που κάποιος ε, είναι τέλειος, ε, δεν ξέρω, εγώ αυτό το φοβάμαι, το να είναι κανείς τόσο τέλειος, αυτό μένα μου προκαλεί τρόμο. Παρακαλώ να πω ότι είμαστε... Θα ήθελα να πω ότι είμαστε τέλειοι, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κάνουμε σφάλματα και προσπαθούμε να διδαχθούμε απαλφά. Επίσης, ε, να σας καθησυχάσω ότι επίσης απολύουμε και κάποιους ανθρώπους, όχι τόσους πολλούς, γιατί είναι μακρά διαδικασία και δεν ανανεώνουμε τις συμβάσεις. Έτσι λοιπόν, τα παίρνουμε όλα αυτά πολύ σοβαρά, θα εξετάζουμε το θέμα της επίδοσης, των πειθαρχικών μέτρων, της παρενόχλησης και με αυτό ασχολείται ο Γενικός και εγώ. Τώρα, για να επανέλθω στις ερωτήσεις σας ε, για την έρευνα στο προσωπικό, δεν είδαμε ιδιαίτερο σύνδεσμο μεταξύ των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής και μιας ένδειξης ότι οι άνθρωποι που νιώθουν άγχος ε, ε, ή μπορεί να εργάζονται περισσότερο, να παθαίνουν burnout. Έτσι λοιπόν, επίσης, το να εργάζεται κανείς στη διπλωματία είναι μια αγχώδης δουλειά και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Θέλουμε οι άνθρωποι να πηγαίνουν και διακοπές, να παίρνουν άδεια. Και λαμβάνουμε όσα μέτρα μπορούμε για να αυξήσουμε την ισορροπία μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματική ζωής, ε, με τηλεεργασία, παραδείγματος χάρη ή με μερική απασχόληση. Αυτά είναι κάποια μέτρα που παίρνουμε μαζί από την Κομισιόν ε, για το προσωπικό στις αντιπροσωπείες. Τώρα είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδεις στην εργασία τους. Αυτό προκύπτει από την έκθεση και περισσότερες κριτικές έχουν να κάνουν με την επικοινωνία, με τη διοίκηση, με την κακή διοίκηση μερικές φορές. Έτσι λοιπόν εργαζόμαστε σε αυτά μαζί με την Κομισιόν για να αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις που προέκυψαν γιατί για πρώτη φορά πέρσι είχαμε μία επισκόπηση που ήταν κοινή για την Κομισιόν και για το προσωπικό της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης ε, που εργάζεται στις υπηρεσίες. Έτσι λοιπόν θα διδαχθούμε από αυτά. Τώρα για την ισορροπία των δύο φύλων. Ναι, προσπαθούμε να προσελκύσουμε γυναίκες και για διοικητικές θέσεις. Έχουμε ένα δίκτυο και συζητάμε πολύ με τους συναδέλφους ε, στην Υπηρεσία Ανθρωπίνων Πόρων όχι μόνο με τα κράτη-μέλη, αλλά και με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Είμαστε και σε ανταγωνισμό με τα κράτη-μέλη. Το ένα τρίτο των ε, βαθμών ε, AD, της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, προέρχεται από τα κράτη-μέλη. Αν δεν προτείνουν γυναίκες και δεν το κάνουν, γιατί και αυτοί έχουν δικό του στόχο και έχουν πολιτικές και έχουν ε, συγκεκριμένο συμφέρον, ανταγωνιζόμαστε με αυτούς. Ε, δεν είναι κάτι εύκολο. Αυτό που θα αλλάξει και θα αλλάξει γιατί έχουμε έναν πληθυσμό που γυράσκει και θα θέσουμε στόχους πρόσληψης ε, νέων γυναικών. Φυσικά θα χρειαστεί χρόνος. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που στην Κομισιόν έχουμε 40% ε, σε διευθυντικές θέσεις στην Κομισιόν. Όμως αυτό ξεκίνησε πριν 20 χρόνια και είχαμε υποχρεωτικό στόχο για τις προσλήψεις ε, γυναικών. Θα χρειαστεί λοιπόν χρόνος επισήμως. Θα χρειαστεί χρόνος έτσι ώστε και οι γυναίκες συνάδελφοι που θα έρχονται από τα κράτη-μέλη να ενδιαφέρονται να έρθουν και στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης για 4-8 χρόνια. Τώρα για τους ασκούμενους. Είχαμε μεγάλες βελτιώσεις χάρη στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του διαμεσολαβητή. Χαιρόμαστε που τώρα μπορούμε να προσφέρουμε τόσο υψηλό αριθμό εγκαταστάσεων άσκησης της αντιπροσωπείες το 2017 ήταν το τελευταίο έτος που δεν χρηματοδοτήσαμε τους ασκούμενους, έπρεπε οι ίδιοι να χρηματοδοτήσουν τον εαυτό τους. Και έχουμε διαφορετική διευθέτηση για τους ασκούμενους στις αντιπροσωπείες. Και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που θέλουμε να τηρήσουμε. Θα μπορούσαμε να μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε γραπτός. Σε ό,τι αφορά τώρα τα θέματα της εμπιστευτικότητας ε, και όλες τις σχετικές ερωτήσεις που θέσατε και το πόσο οργανωνόμαστε. Έχουμε φτάσει στο συνέδριο έξι αντιπροσωπείες ε, και άλλους δύο θα έχουμε του χρόνου. Εγώ ως εκπρόσωπος της διοίκησης δεν έχω λόγο. Είναι η υπηρεσία διαμεσολάβησης που είναι ανεξάρτητη η οποία ασχολείται με το θέμα αυτό και είναι ανεξάρτητη από μένα. Φυσικά, οι συνάδελφοι πρέπει να καταρτίζονται σε πολύ συγκεκριμένα θέματα και ψυχολογική υποστήριξη και πρόληψη των συγκρούσεων. Και έχουμε πολλές περιπτώσεις που έφεραν στην προσοχή μας, το χάρη παρενόχληση ή κάποιες διανέξεις. Βέβαια, είναι καλό σημάδι που οι άνθρωποι τώρα εκφράζονται και υπάρχει μια υπηρεσία, κάποιο αρμόδιο με τον οποίο μπορεί να έρθουν σε επαφή. Γίνεται μια προσπάθεια. Υλοποιούμε και σεμινάρια και τους καλούμε να παρευρεθούν στις Βρυξέλλες. Και είναι πιθανότητα κάτι που διευρύνεται. Όμως δεν μπορούμε φυσικά να αγκάσουμε τους ανθρώπους ε, να γίνουν εμπιστευτικοί σύμβουλοι. Είναι μια απόφαση που αφορά τον καθένα. Και θα σταματήσω εδώ. Και φυσικά μπορούμε να σας δώσουμε γραπτός λεπτομερέστερες απαντήσεις. Gibt's noch weitere Fragen? Δεν ξέρω αν έχετε να κάνετε άλλες ερωτήσεις. Συνάδελφος Κινίτσι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Μογκερίνη που έπρεπε να μας αφήσει γιατί είχε ανηλυμένε υποχρεώσεις στην Ολομέλεια, όπως και τον ε, κύριο Πέτιο Ρούσο για τις παρουσιάσεις τους και ευχαριστώ και σας κύριε που μας δώσατε απαντήσεις στις πολυάρτημες ερωτήσεις. Φυσικά ε, ακούσαμε για μια κατάσταση, είναι πλάκη η υπηρεσία εξωτερικής δράσης σε μια σειρά δραστηριοτήτων σε μια δύσκολη χρονική στιγμή. Υπήρχαν πάρα πολλές προκλήσεις, ε, κλιματική αλλαγή, τρομοκρατία ε, και φυσικά και πάρα πολλές σειράξεις σε διάφορες περιοχές. Και Ακούσαμε και τη δουλειά που κάνατε σε διάφορα επίπεδα και σε ό,τι φορά και το πόσο οργανώνεται η οργανωτική δομή. Τώρα για είναι απαλλαγή. Νομίζω ότι αποτελεί μια ευκαιρία για να γίνει ένας απολογισμός τι έγινε, τι βελτιώθηκε, τα ακούσαμε αυτά, αλλά και τι απομένει προς βελτίωση. Εγώ έχω μια απλή και άμεση ερώτηση. Τι παραμένει να βελτιωθεί κατά την άποψή σας όχι, όχι σε ό,τι αφορά μόνο τις δραστηριότητες, αλλά για την καλύτερη χρήση του προϋπολογισμού της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Τι θα μπορούσαμε ακόμη να βελτιώσουμε, λοιπόν. Ευχαριστώ. Um, thank you very much. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλετε τον κατάλογο αλφαβητικά ή κατά προτεραιότητες, αλλά είναι τόσα πολλά που πρέπει να κάνουμε. Ήδη μας δώσατε πολλά στοιχεία για πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν. Εγώ θα έλεγα, καταρχήν, η ασφάλεια είναι μία από τις μεγάλες μας ανησυχίες. Δεν έχουμε τα μέσα που έχουν οι Ηνωμένε Πολιτείες. για να προστατεύσουμε τις πρεσβείες. Θα πρέπει να συνεργαστούμε περισσότερο με τα κράτη-μέλη. Και για να προστατεύσουμε την πρεσβεία μας, συνήθως ε, προσλαμβάνουμε ακριβές υπηρεσίες ασφαλείας και έχουμε διάφορα ζητήματα, σοβαρότερα ή λιγότερο σοβαρά. Και επίσης ε, βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν την αστυνομία. Αυτή θα ήταν μια ιδέα. Τώρα, το άλλο θέμα είναι η ευελιξία. Έχουμε μια άκαμπτη δομή. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο τη δική μας υπηρεσία, αφορά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και δεν είμαστε αρκετά ε, εύκαμπτη για να αναπτύξουν προσωπικό σε αντιπροσωπή όταν υπάρχει κρίση ή όταν ανακύπτει μια προτεραιότητα. Υπάρχουν στεγανά λοιπόν. Θα ήθελα να εργαστούμε περισσότερο επί διάφορων project και καθηκόντων. Ε, αν προέρχεται κάποιο από τη μία υπηρεσία ή την άλλη αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη ή ένα project να μπορώ να ε, χρησιμοποιήσω τους κατάλληλους ανθρώπους, παραδείγματος χάρη η παραπληροφόρηση. Αναφερθήκαμε σε αυτό και στο θέμα της ασφάλειας. Είναι κάτι που μεγενθύνεται. Δεν θα φύγει και δεν έχουμε την εμπειρογνωσύνη. Ξέρω ότι το Κοινοβούλιο και ορθώς το κάνει και το λάβαμε υπόψη, έχει ζητήσει τη μείωση των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων. Όμως αυτή η εμπειρογνωμοσύνη δεν μπορεί να βρει σε γενικούς διαγωνισμούς. Ε, θα πρέπει ε, να έχουμε ε, έναν εθνικό εμπειρογνώμονα αποσπασμένο ή να έχουμε συμβασιούχους. Επίσης, τώρα με τους συναδέλφους εξετάμε, ζούμε το πώς θα δώσουμε μια διαφορετική υποστήριξη στις αντιπροσωπείες. Θέλουμε ουσιαστικά να αφήσουμε κατά μέρους ε, κάποιες λεπτομέρειες και θέλουμε να επικεντρωθούμε σε θέματα όπως πριν το χάρη οι προμήθειες για την υποστήριξη σε αντιπροσωπείες είχαμε το Περιφερειακό Κέντρο που υποτίθεται ότι θα ήταν ε, το πρώτο από πολλά στην περιοχή. Δεν θα δημιουργήσουμε όμως άλλα τέτοια κέντρα γιατί δεν έχουμε τους πόρους, όμως θέλουμε να βελτιώσουμε επίπεδο της επαγγελματικότητας και αυτό έχει να κάνει με την εικόνα σου και το brand. Αν ε, πας πριν το σχάρι σε μια χώρα και επισκεφτείς μια αντιπροσωπεία θα δεις ότι έχουν διάφορες αίθουσες, ε, σημαίες ε, και Πολλά από αυτά είναι πολύ παλιά γιατί τα κληρονομήσαμε από τα γραφεία συνεργασίας της Κομισιόν. Πολλή δουλειά λοιπόν πρέπει να γίνει και βλέπουμε τι κάνουν πολλά κράτη-μέλη στα Υπουργεία για τις δημόσιες συμβάσεις, υπέρνητος χάρη για τις ε, αποστολές χρησιμοποιούν ε, πάντοτε μία και μόνο εταιρεία και ε, θέλουμε μακροπρόθεσμα να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο προσωπικό να ασχολείται με την πολιτική δουλειά. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Πρόεδρος, ε, νομίζω ότι οι ερωτήσεις ε, του συναδέλφου Κινέα δεν απαντήθηκαν ακόμα, τουλάχιστον όσον αφορά τη Ρωσία. Ίσως ο συνάδελφος Κινέα μπορεί να επαναλάβει, να το επενθυμίσει λιγάκι, γιατί νομίζω ότι εκεί έμεινε κάτι αναπάντητο. Ευχαριστώ. Ναι, είναι θέμα μέσων που διαθέτουμε. Η πρώτη συνάντηση που είχα με το νέο, είπα το εκπρόσωπο, με ρώτησε «Έχεις αρκετό προπολογισμό» Του είπα «Ναι, μένα, αλλά εξαρτάται για την πράγμα». Αν θέλετε να αυξήσουμε την ασφάλεια ή να καταπολεμήσουμε την παραπληροφόρηση, ε, δεν έχουμε τόσο μεγάλους πόρους όπως έχουν μερικές φορές τρίτες χώρες για να φτιάχνουν ψεύτικα προφίλ και να διαδίδουν ψεύτικες ειδήσει. Ε, είπατε ότι είναι αστείο το σχέδιο που έχουμε γιατί έχει πολύ χαμηλό προπολογισμό. Ε, είναι το πρώτο βήμα και θα αυξηθεί αν συμφωνήσουν οι δημοσιονομικές αρχές. Σημαντικό είναι πάντως να το συνδέσουμε με τις διάφορες υπηρεσίες και τους οργανισμούς στις διάφορες χώρες μέλη που καταπολεμούν την παραπληροφόρηση. Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης είναι ήδη κάτι, κυρίως σε περίοδο εκλογών γιατί έτσι μπορούμε, αν μη τι άλλο, να επισημάνουμε την προπαγάνδα που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνική δικτύωση, για παράδειγμα. Οπότε, ναι, είναι, ένα, είναι μια αρχή. Δεν θα σταματήσουμε εδώ. Αν θα τα καταφέρουμε, να αντιμετωπίσουμε τους αντιπάλους μας. Ε, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, δεν ξέρω, πάντως ε, προσπαθούμε. Πρέπει βέβαια να ξέρουμε τι κάνουν και οι άλλοι. Αλλά ήδη αυτά που κάνουμε εμείς είναι σημαντικά. Και ναι, είναι η Task Force της Βρυξέλλης που καταπολεμούν την παραπληροφόρηση, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερο κόσμο και στις αντιπροσωπείες, οι οποίες κινδυνεύουν από τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται η παραπληροφόρηση με συγκεκριμένα επιχειρήματα επιτόπου. Πολύ ωραία. Ε, Κατόπιν τούτου θα ήθελα να δώσω και πάλι το λόγο στον εισηγητή μας αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ τους συναδέλφους. Ε, πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπατε, Τον να ακούσει κανείς ε, άλλες απόψεις. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας και νομίζω ότι θα συνεργαστούμε στενά για τη σύνδεξη της τελικής έκθεσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και σας ε, και τους συναδέλφους σας, γιατί νομίζω ότι είναι απαραίτητο να μιλάμε ανοιχτά. μερικές φορές μπορούμε και εμείς να σας δείξουμε ένα άλλο τρόπο πώς να βλέπετε τα πράγματα, γιατί έχουμε μακρά εμπειρία και θεωρώ ότι είναι καλό και εσείς ε, να μιλάτε για αρνητική εμπειρία. Όλα αυτά μπορούν να βελτιωθούν, γιατί σε τελική ανάλυση ουδής τέλειος. Και ευχαριστώ τους συναδέλφους. Όταν μιλάμε για τα σφάλματα, Κοιτάξτε, ε, στο μέλλον δεν θα εστιάσουμε την προσοχή μας στο ποσοστό σφαλμάτων, αλλά στο πλαίσιο, στο περιεχόμενο, γιατί έτσι μπορεί κανείς να κατανοήσει καλύτερα το ποιο ήταν το πρόβλημα και πώς ακριβώς ε, μπορεί το πρόβλημα αυτό να εξαλειφθεί στο μέλλον. Ε, για μας το σημαντικότερο είναι η γεωγραφική ισορροπία. Ζητώ συγγνώμη και τον προτέρων γι' αυτό, αλλά έτσι θα είναι και εάν κάποιος από εμάς ε, γίνει τελικά εισηγητής για το 2019, ε, θα πούμε θετικά πράγματα για το 2019. Θα αναφέρουμε ότι υπάρχει μικρή πρόοδος, όχι τεράστια πρόοδος, γιατί αν τελικά ήταν ε, δυνατόν να αλλάξει η ισορροπία στο θέμα των δύο φύλων, πόσο μάλλον πολύ πιο εύκολο θα είναι να αλλάξει στο θέμα το γεωγραφικό, γιατί η μεν ισορροπία των δύο φύλων ανάγεται στα τελευταία 100 χρόνια, ενώ το γεωγραφικό στα τελευταία 15 χρόνια. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους, ε, το ελεγκτικό συνέδριο, ε, τον κύριο Ρούσο, ο οποίος ε, έγραψε αυτή την έκθεση, ήρθε σε εμά ε, στο Στρασβούργο, αλλά να ευχαριστώ και εσά θερμά, κύριε Γενική Γραμματέα, για την ε, εξαιρετική συνεργασία και σας παρακαλώ να διαβιβάσετε τις ευχές μας στην κυρία Μογκερίνη, να τις διαβιβάσετε ότι σεβόμεθα τόσο τη δική της ε, προσωπική εργασία αλλά και αυτή των συνεργατών τη ε, στην υπηρεσία εξωτερική δράση. Τώρα υπάρχει ένα προβληματάκι θα το έλεγα. Ε, δεν έχει έρθει ο Επίτροπος. Α, μισό λεπτό λέει η πρόεδρο, έκανα λάθος, δεν χάσαμε Επίτροπο, ήρθε ο Επίτροπος. Αγαπητέ Επίτροπε, κύριε Μίμικα, ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που ήρθατε σήμερα εδώ, μπορώ να σας καλωσορίσω και χαίρομαι επίσης ε, που από πλευράς ε, ελεκτικού συνεδρίου έχουμε τον κύριο Τομέμ Κουρούσα και ως μέλος του Ελεκτικού συνεδρίου θα μας ενημερώσει, θα προβεί στην πρώτη ανάλυση του ελεγκτικού συνεδρίου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, είναι μεγάλη τιμή για μένα που μπορώ και βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή σα για να σα παρουσιάσω στα πλαίσια τη διαδικασία απαλλαγή τα αποτελέσματα του έργου του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την κατηγορία 4, μια συνολική Ευρώπη τη ετήσια έκθεσή μα για το 2018. Αυτό το πλαίσιο δαπανών αφορά τι δαπάνε εξωτερική πολιτική, την πρόθεση των αξιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη στήριξη των υποψηφίων χωρών, όπω επίση και τη συνεργασία στην ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια συνολικά ανά τον κόσμο. Το 2018 λοιπόν. Οι δαπάνες που ελέγξαμε εμείς ήταν 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε αντίθεση με άλλα κεφάλαια τη ετήσιας εκθεσή μας, δεν κάνουμε μια ειδική αξιολόγηση τη πολιτική αυτή. Το δικό μας έργο ήταν να ελέγξουμε ένα δείγμα 58 συναλλαγών, όπου διαπιστώσαμε σε 11 περιπτώσεις σφάλματα. Από αυτές τις 11 συναλλαγέ με σφάλμα, 5 εκφράστηκαν ποσοτικά και συζητήσαμε τις νομικές επιπτώσεις. Επίσης, το ελεγκτικό συνέδριο εντόπισε μία περίπτωση δαπανών που συμπεριλαμβάνονται στην δήλωση δαπανών. Για παράδειγμα, στα πλαίσια ενό ε, σχεδίου που ελέγξαμε, εντοπίσαμε ανάμεσα στα διάφορα δικαιολογητικά δαπάνες ε, ταξιδιών που δεν είχαν επιδοτηθεί επίσης και μία περίπτωση όπου δεν σεβαστήκαμε τις διαδικασίες ε, διαγωνισμών. Επίσης έχουμε συμπεριλάβει στην έκθεσή μας και ένα παράδειγμα αποτελεσματικών ελέγχων που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε παραδείγματα στην έκθεσή μας με πολλές καλές πρακτικές από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, η κατηγορία «Μια συνολική Ευρώπη» Ε, είναι κάτι το οποίο χειρίζονται διάφορες γενικές διευθύνσεις. Η ΔΕΦΚΟ, η Γενική Διεύθυνση για τη Συνεργασία για την Ανάπτυξη, η ΝΙΡ, η Γενική Διεύθυνση για τις ε, Πολιτικές Διεύρυνσης και Γειτονίας, η Γενική Διεύθυνση επίσης Προστασίας των Πολιτών και Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Όπως επίσης ε, συμμετέχουν και υπηρεσίε που ασχολούνται με τα μέσα εξωτερικής πολιτικής αλλά και με τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πάνω από 150 χώρες. Επίσης, έμεσα οι χώρες δικαιούχοι και διάφοροι διεθνείς οργανισμοί μπορούν επίσης να συμμετέχουν στην διαχείριση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας εδώ Επίσης, τι δυσκολίες ε, που αντιμετωπίσαμε φέτος προκειμένου να πετύχουμε έγκαιρα τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να κάνουμε τη δουλειά μας σε διάφορες ε, περιπτώσεις από την UNICEF αλλά και από το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφοδότησης στο ΙΕ. Η έλλειψη συνεργασίας προκειμένου να μα φτάσουν ε, τα διάφορα δικαιολογητικά ή που χρειαζόμαστε επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό τον σχεδιασμό των δικών μας ελέγχων. Και έτσι προβήκαμε σε σύσταση προς αυτή την κατεύθυνση. Πέρα λοιπόν από τον έλεγχο των συναλλαγών που χρησιμεύουν για να αποφασίσουμε ποιο είναι το ποσοστό σφάλματος, η έκθεσή μας αναλύει και το, σφάλμα, το επίπεδο σφάλματος στην περίπτωση των πολιτικών γειτονίες και διεύρυνσης. Και ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των γενικών διευθύνσεων από την ΤΕΦΚΟ και την ΕΚΟ επίσης εξετάστηκαν από εμά. Το 2018 λοιπόν όσον αφορά την DGNIR έγινε μελέτη για το σφάλμα που ανατέθηκε σε μια εξωτερική υπηρεσία και το λεκτικό συνέδριο ε, κατέληξε στο ότι διπλασιάστηκαν οι περιπτώσεις όπου υπάρχει πλήρης ε, εμπιστοσύνη στα καλά αποτελέσματα. Και επίσης επαληθεύτηκε το ότι το έργο αυτό από τους εξωτερικούς ελεγκτές έγινε σωστά. Όσον αφορά τώρα τη δυνατότητα διόρθωσης του σφάλματος από πλευρά της Γενικής Διεύθυνσης για την Προστασία του Πολίτη και Ανθρωπιστική Βοήθεια, πέρα από τις προσπάθειες που έγινε να μην υπολογιστούν η προχρηματοδότηση και ακυρωμένες πληρωμές, εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι, η... ότι τα ποσά τα οποία αναφέρονται είναι υπερεκτιμημένα. Επίση, προσπαθήσαμε να ελέγξουμε την νομιμότητα και την κανονικότητα της διαχείρισης και το ελεγκτικό συνέδριο ε, κατέληξε σε 15 περιπτώσεις που δεν ήταν σωστές και κάναμε ελέγχους σε θέματα απόδοσης επιτόπου στην Ουκρανία, την Αλγερία, την ε, Βοσνία, Ριζεγοβίνη και το Λάος. Εκτός από μία περίπτωση όλα τα σχέδια τα οποία εξετάστηκαν είχαν δείκτες σαφού σαφούς απόδοσης και καταλληλότητας. Επίσης τα πλαίσια τα καλά διαρθρωμένα και οι στόχοι ήταν ρεαλιστικοί και βιώσιμοι. Σε αυτά τα πλαίσια, επίση, το Ελεκτικό Συνέδριο κατέληξε σε τρει συστάσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, η πρώτη σύσταση, στην οποία αναφέρθηκα και νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να ενισχύσει την υποχρέωση των διεθνών οργανισμών να μεταφέρουν στο ελεγκτικό συνέδριο οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία η οποία βοηθάει ώστε να επιτελέσουμε και εμείς το έργο μας. Δεύτερον, συστήσαμε να υιοθετηθούν μέτρα προκειμένου να προσαρμοστεί η μεθοδολογία της ε, μελέτης για το υπόλοιπο σφάλματος, το υπολοιπόμενο σφάλμα, έτσι ώστε να περιοριστούν οι περιπτώσεις που βασίζονται σε πλήρη εμπιστοσύνη στο έργο τρίτων από άλλους δηλαδή ελεγκτές. Και τέλος, η σύστασή μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει τον υπολογισμό που γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση Προστασίας των Πολιτών και Ανθρωπιστικής Βοήθειας για την ικανότητα διόρθωσης όσον αφορά το 2019, αφαιρώντας ε, τις επιστροφές από την ε, μικρότερη χρησιμοποίηση των ποσών. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεργασία της με το ελεγκτικό συνέδριο και για το θετικό κλίμα συνεργασίας που υπήρξε μεταξύ μας όλα αυτά τα χρόνια. Ώστε να καταλήξουμε και εμείς αυτή την ετήσια έκθεση που σας παρουσιάζουμε σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή ερώτηση έχετε. Ευχαριστώ. Καταρχάς ε, να ευχαριστήσω θερμά για αυτή την ε, ακριβή παρουσίασή σας και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Μίμικα. Σας ευχαριστώ πολύ, ε, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Πριν λοιπόν ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης ε, και για τις λεπτομερείς παρατηρήσεις σχετικά με τις εξωτερικές μας παρεμβάσεις, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον, την, την πρόεδρο της Επιτροπής και η συγγετρία την κυρία Χολμάια που με κάλεσε σε αυτή τη συνεδρίαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παίρνει πολύ σοβαρά τη δουλειά του ελεγκτικού συνεδρίου. Συγκεκριμένα το 2018 για άλλη μια φορά εφαρμόσαμε τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου προχωρήσαμε με σύνεση, με διαφοροποιημένη ανάλυση για τα ποσοστά ασφάλματος ε, και, για, και με σαφείς δράσεις άμβλυνσης για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις αδυναμίες που παρουσίασε το ελεγκτικό συνέδριο. Επειδή το ελεγκτικό συνέδριο παρουσίασε μόνο ένα ποσοστό ασφάλματος για το σύνολο του ευρωπαϊκού προπολογισμού και δεν υπάρχουν πλέον εκτιμήσεις ε, κατά κεφάλαιο, ε, το θέμα του ποσοστού σφάλματος θα το αναφέρω όταν θα έρθω στην απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Και φτάνω τώρα στην δεύτερη πρόκληση, δηλαδή του πώς οι πολιτικές και οι πόροι μπορούν να μετατραπούν σε ορατά αποτελέσματα. Ε, εγώ εξακολουθώ να είμαι δεσμευμένος ε, τον ε, έλεγχο και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ε, να την κάνω όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική. Πέρα από αυτά που δαπανάμε θα πρέπει να εξετάζουμε και τους στόχους, τους στόχους των προγραμμάτων που, έχει, που έχουν προκύψει. Ξεκινάμε με την υποστήριξη του προϋπολογισμού που μας ε, επιτρέπει ε, στο διάλογο υψηλού επίπεδου, μας επιτρέπει να έχουμε διάλογο υψηλού επίπεδου, διαρθρωμένο διάλογο με τις γειτονικέ χώρες για θέματα που είναι καθοριστική σημασία για την ανάπτυξή τους, παραδείγματος χάρη χρηματοδότηση των δημόσιων δαπανών, διαφθορά, ποιότητα των πολιτικών και μακροοικονομική σταθερότητα. Ε, θεωρώ ότι είναι επένδυση αυτό στα συστήματα των εταίρων μας για να μεταρρυθμιστεί η διοίκηση, να προσφέρονται καλύτερες υπηρεσίες, οι κυβερνήσεις να είναι περισσότερο ε, αποτελεσματικές στη λογοδεσία και στη διαχείριση, να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη διαφθορά. Κατά την άποψή μου αυτό αποδίδει. Ίσως η πρόοδος ε, να μην είναι ακριβώς ίδια σε όλες τις χώρες, αλλά σε γενικές γραμμές οι τάσεις που επικρατούν λένε πολλά από μόνες τους. Ε, η αξιολόγηση των προγραμμάτων υποστήριξη προπολογισμών. Οι αξιολογήσει αυτέ ε, επιβεβαιώνουν αυτά τα οποία σα είπα. Η υποστήριξη των προπολογισμών διασφαλίζει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και είναι ο καλύτερο τρόπο για να στηρίζεται ο διάλογο με του εταίρου μα. Οι χώρε εταίροι, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, η κοινωνία των πολιτών, οι υπηρεσίε αξιολόγηση όλοι έχουν καταθέσει ότι η υποστήριξη των προπολογισμών προπολογισμών λειτουργεί πολύ καλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσβλέπει ε, στο να ε, πουλήσει, να επικοινωνήσει προς τα έξω αυτά τα καλά αποτελέσματα. Επίσης έχουμε στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς, προφανώς με τα Ηνωμένα Έθνη, την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και αυτό για να δοθεί μεγαλύτερη υποστήριξη και να υπάρχει μεγαλύτερη κινητοποίηση γενικότερα ε, στην υποστήριξη προπλογισμών. Συγκεντρώνοντας πόρους και μοχλεύοντας εθνικούς πόρους ε, για να γίνεται καλύτερη χρήση της τεχνογνωσίας μας σε διάφορους τομείς ή σε συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό ακριβώς έλαβε χώρα. Σε άλλα θέματα έχουμε πρόοδο στην εφαρμογή των τεσσάρων καταπιστευματικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χάρη αυτών η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε παρουσία και έχει καταδείξει καθοδηγητικό ρόλο στο συντονισμό των κρατών μελών και άλλων δωρητών. Τα καταπιστευματικά τα ταμεία μας επέτρεψαν επίσης να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και ε, να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα συγκεντρώνοντας πόρους ε, και χρησιμοποιώντας διαδικασίες ταχύτερης έγκρισης και εφαρμογής και ε, διασφαλίζοντας την κατάργηση των αποκλεισμών. Η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό είναι πολύ αποτελεσματικό. Έχουμε επίσης σημειώσει αρκετή πρόοδο στην εφαρμογή, στην εκτέλεση του προγράμματος εξωτερικών επενδύσεων 1,5 ευρώ έχουν εκταμιευτεί ε, σε 28 συμβάσεις ε, με στόχο να μοχλεύσουν πάνω από 17 δις ιδιωτικών επενδύσεων μέσα από, την, ε, από διευκολύνσεις και την μείωση των κινδύνων. Σε αρχές του μήνα υπέγραψα δύο τέτοιες συμφωνίες. Επιπλέον πάνω από 2,5 δις ευρώ είναι υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκταμιεύτηκε σε blending παρεμβάσεις ε, στην Αφρική, στη γειτονιά μας ή ξεμπλοκάροντας επενδύσεις 24 δις ευρώ σε ελπιδοφόρους τομείς της οικονομίας όπως είναι μεταφορές, η βιώσιμη οικονομία αλλά και άλλα, άλλοι τομείς όπως η βιώσιμη γεωργία. Τέλος, έγιναν διαπραγματεύσεις για το ε, εργαλείο εξωτερικής, εξωτερικών επενδύσεων από το 21 μέχρι το 27 στο επόμενο πουδουπού γίνονται αυτές οι διαπραγματεύσεις. Η τρίτη, ο τρίτος τριμερής διάλογος θα λάβει η χώρα τον 8, μάλλον με έλαβε χώρα τον Οκτώβριο και αυτό ήταν μια πολύ καλή αρχή. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για να ξεκινήσει η πρόοδο σε αυτό το θέμα, να εγκριθεί έγκαιρα και να αρχίσει να εφαρμόζεται τον Ιανουάριο του 2021. Γνωρίζω ότι ε, το Κοινοβούλιο συμμερίζεται το δικό μας στόχο που είναι να μεγιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό να γίνει προτεραιότητα για την επόμενη οικονομική περίοδο. Γι' αυτό ε, πραγματικά προσβλέπω στη συνεργασία με εσά. Επανέρχομαι ε, στις, ε, στην απαλλαγή αυτού του έτους. Ε, δύο επιφυλάξει έχουμε στην τήσια έκθεσή μας για το 2018. Πρώτον, έπρεπε να εκφράσουμε μια, να στηρίξουμε την επιφύλαξη που αφορά στις άμεσες επιχορηγήσεις. DG DEFCO δόθηκαν στη DG NIA το 2018. Η δεύτερη επιφύλαξή μας έχει σχέση με τη διαχείριση των ταμείων από την Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής. Έπρεπε να διατηρήσουμε αυτή την επιφύλαξη γιατί εξαρτάται από το αποτέλεσμα της νέας αξιολόγησης αυτού του θεσμού που θα ολοκληρωθεί στο τέλος αυτού του έτους. Αν τα αποτελέσματα είναι θετικά, υπάρχει πιθανότητα να αρθεί αυτή η επιφύλαξη κατά το επόμενο έτος. Αξιότιμα μέλη, η δική μας η προσοχή είναι και θα είναι στο να επιτυγχάνουμε τα μέγιστα αποτελέσματα και την πλήρη εκμετάλλευση, την βέλτιστη εκμετάλλευση των κονδυλίων μας. Το οφείλουμε αυτό στους προλογούμενούς μας και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους ανά τον κόσμο που ε, αποφελούνται από τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με άλλες χώρες για αναπτυξιακά θέματα. Και αν ε, μας στηρίξετε θα συνεχίσουμε να κατευθυνόμεθα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, νομίζω τώρα υπάρχει κάποια, κάποιο μπέρδεμα. Ε, διότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, η συνάδελφος βλέπω χαμογελάει, απευθύνομαι ε, στη συνάδελφο στο συνάδελφο, μάλλον στη συνάδελφο, να ξεκινήσει εσύ με το EDF ε, και μετά εγώ θα συνεχίσω με το ΕΦΚΟ ε, και δεν θα χρειαστεί να ε, ξαναεπέμβει ο Επίτροπος. Θα τα χειριστούμε πολύ καλύτερα με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, εσύ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Βέβαια, αν συμφωνεί και ο Επίτροπος ή με θέλει το μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου να πει κάτι για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Ε, κάπως και εγώ τώρα ε, είμαι σε δύσκολη θέση πρέπει να σας πω. Ε, να δώσουμε καλύτερα το λόγο καταρχήν στον εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου και μετά εμείς για να μην τα μπερδέψουμε. Και αφού τα μπερδέψαμε ας παραμείνουμε σε αυτό το μπέρδεμα λέει η Πρόεδρος. Κυρία Πρόεδρε, θα σας παρουσιάσω με ικανοποίηση την έκθεση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης στο οικονομικό έτος 2018 ελέγξαμε 4 ε, εκατομμύρια 100 εκατομμύρια ευρώ. Ε, Όπω ε, ξέρετε, τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξη αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέχει ενίσχυση στην αναπτυξιακή συνεργασία. Σύμφωνα με την άποψή μα, οι αιτήσιοι λογαριασμοί του 8ου, 1ου, 10ου, 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξη το 2018 παρουσιάζουν πιστά σε όλες τις σημαντικές τους πτυχές στην οικονομική τους κατάσταση στις 21η Δεκεμβρίου και τα αποτελέσματα των συναλλαγών των ταμιωκών ροών και οι αλλαγές ε, των, του καθαρού πνευματικού. Επίσης αντικατοπτρίζεται τα έσοδα ε, είναι νόμιμα και κανονικά. Σε ό,τι αφορά τις ε, δαπάνες, ε, οι λογαριασμοί έχουν ένα ποσοστό σφάλματος 5,2% ανώτερο από το όριο σημαντικότητας που θέτει η μεθοδολογία μας που είναι 2%. Αυτό μας οδηγεί στο να εκδώσουμε μια αρνητική γνώμη σε σχέση με την ομότητα και κανονικότητα των δαπανών αυτών των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης. Το 2018 ελέγξαμε ένα δείγμα 125 συναλλαγών. Από αυτές οι 51 παρουσίαζαν σφάλματα από τα οποία τα 39 είχαν δημοσιονομικό αντίκτυπο. Το μεγαλύτερο μέρος των σφαλμάτων έγιναν ε, λόγω της έλλειψης των κατάλληλων δικαιολογητικών εγγράφων, λόγω ε, μη σεβασμού των κανόνων ε, στις δημόσιες συμβάσεις και από την αποδοχή δαπανών μη επιλέξιμων. Είδαμε ότι σε ορισμένε περιπτώσει όπου βρήκαμε σφάλματα, η Επιτροπή διέθετε επαρκεί πληροφορίε ε, στου ε, φακέλου δαπανών, ε, έτσι ώστε να μπορούσε να τα έχει αποφύγει, να τα διορθώσει πριν να δεκτεί την πληρωμή. Αν είχε χρησιμοποιηθεί καταλήλωση πληροφορίες, το εκτιμόμενο επίπεδο σφάλματος στις δαπάνες των ταμείων θα ήταν 1,2% χαμηλότερο. Όπως ε, σας είπα στην ε, προηγούμενη ε, ομιλία μου σε σχέση με την παγκόσμια Ευρώπη, στην περίπτωση του ΕΤΑ είχαμε κάποια προβλήματα λόγω έλλειψης συνεργασίας με κάποιους διεθνούς οργανισμούς και αυτό μας οδήγησε στο να διατυπώσουμε στην Κομισιόν μία παρόμοια σύσταση με αυτή που έχουμε στην ετήσια έκθεση σε σχέση με την ε, ανάλυση που υλοποιήσαμε για την ε, μελέτη για το υπολοιματικό ποσοστό λάθους ε, από την ΓΑΜΑ που ζητήθηκε από την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ τονίσαμε κάποιους περιορισμούς στην μεθοδολογία για τον υπολογισμό αυτού του ποσοστού σφάλματος. Καταρχήν, τον μικρό αριθμό των ελέγχων που υλοποιούνται επί τόπου, το ότι οι έλεγχοι που υλοποιούνται σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις δεν είναι πλήρης και τέλος τα συστήματα για την εκτίμηση των υπολογισμών των σφαλμάτων. Γι' αυτό συστήνουμε στην Κομισιόν να βελτιώσουμε τη μεθοδολογία και το εγχειρίδιο της ε, μελέτης σε ό,τι αφορά το υπολοιπόμενο ποσοστό σφάλματος. Στις ε, διάφορες επισκέψεις και ελέγχους που υλοποιήσαμε επί τόπου, οι ελεγκτές μας εντόπισαν περιπτώσεις αποτελεσματικής ε, χρήσης ε, των αγαθών και των εγκαταστάσεων ε, που έχουν αποκτηθεί στα πλαίσια των έργων που ελέγξαμε. Έχουμε παραδείγματα βαλτιστών πρακτικών, όμως επίσης βρήκαμε καταστάσεις όπου η αποτελεσματικότητα της δράσης δεν ήταν προφανής ή υπήρχαν αμφιβολίες σε σχέση με τη βιωσιμότητα των ε, έργων που υλοποιούνται με ευρωπαϊκά κονδύλια. Όπως σας είπα, μια λεπτομερέστερη εξήγηση και λεπτομερέστερα παραδείγματα θα βρείτε στην έκθεση που μόλις σας παρουσίασα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή αμφιβολία μπορεί να έχετε. Και εμεί σα ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, από ό,τι άκουσα και είδα, ο κύριο Μιμίκα ε, θέλει να πει κάτι επιπρόσθετα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Α μιλήσει λοιπόν τώρα ο Μήτροπο και μετά α μιλήσουμε οι δυο μα. Στην αρχή, σα είπα, κάπω μπερδευτήκαμε γιατί υπήρξε σύγχυση με την ΤΕΦΚΟ και το EDF, αλλά εν πάση περιπτώσει, παρακαλώ, Επίτροπος. Ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο που μας παρουσίασε την ετήσια έκθεση για το Ευρωπαϊκά Ταμείο Ανάπτυξη. Καταρχήν ε, να επικεντρωθώ σε θέματα που αφορούν ε, το ΕΤΑ. Και πάλι ευγνωμονούμε το Ελεγκτικό Συνέδριο για τις συστάσεις και για το έργο του συνεχίζει να διέπει και να καθοδηγεί τις συνεχείς προσπάθειες της Κομισιόν να βελτιώσει το σύστημα ελέγχου. Το ποσοστό σφάλματος που μέτρησε το συνέδριο για το ΕΤ αυξήθηκε το 2018 παρόλο που δεν είχε αλλάξει η προσέγγιση μας. Η αύξηση αυτή αποτελεί ουσιαστικά μία διακείμενση παρά μία στατιστική τάση προς τα πάνω. Συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε το σχέδιο δράση μας ε, για να απλοποιήσουμε και να αποσαφηνίσουμε του σχετικούς κανόνες και διαδικασίες ε, και ε, να παρέχουμε περισσότερη κατάρτιση στο προσωπικό μας και να έχουμε καλύτερο έλεγχο για να μειώσουμε το ποσοστό σφάλματος τα επόμενα έτη. Επίση, θα προσέξετε ότι το Νεκτικό Συνέδριο στην ετήσια εκθεσή του για τα ΕΤΑ αναφερθήκε σε ε, κάποια έλλειψη συνεργασία από τους διεθνεί οργανισμού. Είναι πράγματι λυπηρό και πιθανότατα λόγω των στενών προθεσμιών που έπρεπε να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Η Κομισιόν θα βάλει τη δυνατά τη για να βελτιώσει τη συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς και να βοηθήσει να εξομαλυνθεί η διαδικασία ελέγχου. Τα καλά νέα ε, είναι ότι το επαγγελματικό ποσοστό φαρματός για τις δραστηριότητε της ΓΔΕΦΚΟ μειώθηκαν περαιτέρω το 2018. Το ε, εκτιμήθη Είναι πιο υψηλό το ποσοστό φάλματο ε, που εκτιμήθηκε για το ΕΤΑ από το υπολοιματικό ποσοστό φαλματό και αυτό είναι κανονικό. Τα δύο ποσοστά φαλματό εξυπηρετούν διαφορετικού σκοπού και δεν μετράνε τα ίδια πράγματα. Το ελεκτικό συνέδριο ε, και το σχετικό του που καλύπτει τις συμβάσεις ε, του ΕΤΑ ορίζεται στην αναλογία του ποσού των μη επιλέξιμων δαπανών ε, σε σχέση με το συνολικό ποσοστό των πληρωμών, ποσό των πληρωμών που υλοποιήθηκαν το συγκεκριμένο έτο, καθώς οι συναλλαγές που αναλύθηκαν από το ελεκτικό συνέδριο κυρίω αφορούν τρέχουσε συμβάσεις, το ποσοστό σφάλματος του συνεδρίου αφορά περισσότερο τις πληρωμές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω ελέγχων επαληθεύσεων, εσωτερικών ελέγχων, εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να διορθώσει ως ένα βαθμό τα σφάλματα που σχετίζονται με αυτές τις συναλλαγές. Το υπολοιματικό ποσοστό λάθος ε, που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της ΓΑΜΑ εκτιμά το ποσοστό φάσματος που παραμένει μη ανιχνεύσιμο δυνάμει αφού έχουν εξαντληθεί όλες οι πιθανότητες για την ε, αποκάλυψή του. Έτσι λοιπόν το υψηλότερο ποσοστό φάσματος ε, στο οποίο αναφέρθηκε το συνέδριο, μας δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να διορθώσει τα σφάλματα πριν να κλείσουν οι συμβάσεις οποιαδήποτε αξιολόγηση για το πώς υλοποιούνται οι συναλλαγές των ΕΤΑ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το επικίνδυνο και πολύ πλοκοπλαίσιο στο οποίο λειτουργούν. Όμως, όπως είπα νωρίτερα, πάντοτε μπορούμε να τα πάμε καλύτερα. Επομένως, ε, κάνουμε συγκεκριμένες δράσεις για να εφαρμόσουμε τις συστάσεις του λεκτικού Συνεδρίου. Οι προσπάθειες αυτές αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και συνδέονται φυσικά με το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο της σχέσης μας ε, με τις ε, χώρες ΑΚΕ να είμαι σαφής. Θα πρέπει λοιπόν να διορθώσουμε το πλαίσιο μετά το κοτονού. Αυτό είναι ζωτικό για να μεταφορμόσουμε τη σημερινή εταιρική σχέση σε μια, ένα πιο μοντέρνο πολιτικό πλαίσιο που να πετυχαίνει τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με την Αφρική, είμαι πεπισμένος ότι η Συμμαχία Αφρικής Ευρώπης για, τη βιώσιμη, ε, για τις επενδύσεις και τις εργασίες είναι σημαντικό ορόσημο για μια ισχυρότερη οικονομική σύμπραξη που θα ωφελεί και τις δύο υπήρους μας και τους πολίτες μας βοηθά στο να υπάρχουν μεγαλύτερε επενδύσει στην ευτική, να δημιουργηθούν θέσει εργασία και να επενδύσουμε στην παιδεία και στι δεξιότητε. Σε ό,τι αφορά τον επιχειρησιακό αντίκτυπο των καταπιστευτικών ε, ε, ε, το Trust Fund για την Αφρική είναι αποτελεσματικό εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στο Σαχέλ, στη λίμνη του Τσάτ, στο κέρας της Αφρικής ε, και αλλού. Επίσης, το Trust Fund του Μπακού έχει δείξει τα ωφέλη του γεφυρώνοντας το κενό μεταξύ ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών δράσεων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία για να εξυπηρετήσουμε το πολιτικό όραμα της συμφωνίας μετά το Κοτονού και έχοντας ακούσει τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε προωθήσει μια πρόταση για να συμπεριλάβουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη στο Γενικό Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κοινοβούλιο, επομένω, θα και τις αρμοδιότητες ελέγχου του και επί των ποσών αλλά και επί το πώς δαπανώνται τα ποσά από τους εταίρους ΑΚΕ. Πιστεύω ότι αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη συνοχή και σε μια μεγαλύτερη έμφαση εν τέλει στα αποτελέσματα και τις επιδόσεις. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, σας επικεντρωθούμε στο να καταστήσουμε τη συνεργασία μας στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξη ώστε δυνατόν πιο αποτελεσματική. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή σας και την επικοδομητική σας συμβολή. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Τώρα λοιπόν εμείς οι δύο συγγήτρες, οι κυρία Ριβάζη και εγώ θα λάβουμε το λόγο γιατί έχουμε περίπου τους ίδιους και συγγητές ε, και για τις δύο εκθέσεις ε, και έτσι θα τα, τα φέρουμε κάπως να ε, μιλήσουμε μέσα στο χρονικό πλαίσιο που προβλέπετε. Και θα ήθελα καταρχήν να δώσω το λόγο στη συνάδελφο κυρία Ριβάζη για να μιλήσει για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Μιμίτσα. Έτσι καλώς γνωριστήκαμε και στην προηγούμενη θητεία. Και ευχαριστώ και το ελεγκτικό συνέδριο. Γιατί είναι καλό να έχουμε ένα ελεγκτικό συνέδριο το οποίο να αναλύει τα αποτελέσματα. Τώρα, θέλω να πω στους συναδέρφους πάντως ότι αυτός ο προπολογισμό του ΦΕΔ είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από τα κράτη-μέλη, είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είναι απόλυτα συνεπής, είναι 74 δισεκατομμύρια. Και είμαστε οι πρώτοι δωρητές παγκοσμίω όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια. Και θα δείτε ότι θεωρώ πως η προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως δεν είναι στο ύψος αυτής της προσφοράς. Και υπάρχουν γενικές διευθύνσει που θα έπρεπε να ζητάνε περισσότερα όσον αφορά την προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξέρετε και στη Γαλλία το έχω αυτό το πρόβλημα έτσι και πάντα τα λέω και φωνάζω ότι δεν είναι γνωστό το τι χρηματοδότηση κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν πάση περιπτώσει. Ο πρώτο στόχο τη δημόσια βοήθεια για την απτυξιακή βοήθεια είναι τελικά η μείωση αλλά και η εξάλληψη πλήρω τη φτώχεια. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο της αναπτυξιακής βοήθειας. Και γιατί το αναφέρω αυτό, γιατί διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια κάπως ανησυχητική τάση όσον αφορά το 11ο ΦΕΔ, που έχει να κάνει με την μετανάστευση και την ασφάλεια, που τελικά απομακρύνεται από τον βασικό στόχο που είναι η εξάλληψη της ε, φτώχειας. δεν πρέπει να παίρνουμε κονδύλια από την εξάλληψη της φτώχειας για τη μετανάστευση. Έπειτα έχουμε τη λήξη της Συμφωνίας Κοτονού το Φεβρουάριο του 2020. Οπότε το τι θα γίνει μετά ε, το Κοτονού αυτό είναι που έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα πρέπει να το σκεφτούμε πολύ. Και κάτι άλλο εισαγωγικά που θέλω να πω είναι το εξή. Ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο αλλά και η Κομισιόν, συμφωνούμε μεταξύ μας αυτό, το ΦΕΔ να ενταχθεί στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Γιατί βλέπετε, θα ψηφίσουμε, θα ψηφίσουμε υπέρ της απαλλαγής, εντάξει, αλλά εμείς, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως βλέπετε, ε, στον προϋπολογισμό μας ενδιαφέρει να υπάρχει το ΦΕΝΤΕ, δεν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία. Λοιπόν, δεν θα επανέλθω στο ελεγκτικό συνέδριο, αλλά στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διατυπώθηκαν στην απαλλαγή του 2017. Ε, σας υποβάλαμε ερωτήσεις, αναλύσαμε τις απαντήσεις σας και εδώ θέλω να προσθέσω κάποια στοιχεία σε σχέση με τις βασικές μας συστάσεις. Πρώτον, υπάρχει μια διορθωμένη αξιολόγηση των δραστηριοτήτων ΟΦΕΔ και στα αποτελέσματα όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και ε, τα δικαιώματα. Εγώ εδώ και 40 χρόνια ασχολούμαι με την Αφρική. Μα καταλαβαίνετε πόσα πολλά χρήματα δίνουμε και όταν λέμε πώς έχουν εξελιχθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα ή το περιβάλλον στην Αφρική, δεν υπάρχει διαρθρωμένη αξιολόγηση. Και αυτό είναι ένα κενό που πρέπει να καλυφθεί. Να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε, να εντοπίσουμε τα αποτελέσματα, να τα συνδέουμε με συγκεκριμένους στόχους. Λοιπόν, εδώ η Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ έχει μια μεγάλη πρόκληση απέναντί της. Έπειτα, για τις άμεσες ενισχύσεις. Πρόκειται για μεταφορά ουσιαστικών ποσών στην χώρα δικαιούχο. Υπέρ της λύσης συγκεκριμένων και τομιακών προβλημάτων με τη βοήθεια μάλιστα και της τεχνικής αρρωγής. Διάβασα την απάντησή σας και ανησυχώ για την χρήση των κονδυλίων αυτών που μεταφέρονται, διότι συγχωνεύονται με τα κονδύλια από τις χώρες εταίρους, άρα δεν ξέρουμε τι γίνεται με αυτά, ιδίως στις χώρες όπου δεν υπάρχει δημοκρατία, έλεγχος κτλ. Και ωραία η δημοσιονομική στήριξη, γιατί μόνο η Ευρώπη την προσφέρει, δεν είναι ούτε Κινέζοι, ούτε άλλες χώρες που το κάνουν. Όμως πιστεύω ότι δεν παρακολουθούμε τι γίνεται με τα κονδύλια αυτά. Και βλέπετε, μπορεί κάποιος να τα βάλει μαζί μας και να μας πει, μα τελικά που πάνε αυτά τα χρήματα. Γι' αυτό λοιπόν και σας ζητώ. Και θεωρώ ότι είναι καλύτερο να βελτιωθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός όσον αφορά τη χώρα δικαιούχου για να μην υπάρχει διαφθορά και όντω να πηγαίνουν τα χρήματα στον προορισμό τους. Έχω και άλλα πράγματα να πω έτσι. Λοιπόν, προβολή της Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνουμε τόσα πολλά χρήματα. Και τελικά οι ίδιοι οι διεθνείς οργανισμοί δεν βοηθάνε σε αυτή την προβολή. Εδώ πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση. Πώς. Πρέπει να ολοκληρώσετε, λέει ο Πρόεδρος. Επιτρέψτε μου δύο λεπτά ακόμα. Καλά, ένα λεπτό. Για τα κατεπιστευματικά ταμεία. Υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα που πηγαίνουν εκεί για την ασφάλεια και τη μετανάστευση. Και εδώ πέρα υπάρχει στρέβλωση στο στόχο του ΦΕΔ τελικά. Και το τελευταίο παράδειγμα είναι η Ερυθρέα. Ήρθανε μη κυβερνητικέ οργανώσεις να με δουν για να μου πούνε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε υπογράψει μια σύμβαση 20 σκατομμυρίων και εσείς δέχεστε ότι η εταιρεία της Ερυθρέας ε, παίρνει κόσμο από την ε, χώρα που σημαίνει ότι βασικά πρόκειται για καταναγκαστική εργασία. Μα πώς θα δικαιολογήσουμε να χτίζει δρόμους στην Ερυθρέα η Ευρωπαϊκή Ένωση με καταναγκαστική εργασία. Πώς σας φαίνεται αυτό. Δεν αισθάνομαι εγώ καλά. Έτσι, να ξέρετε. Και θέλω απαντήσει από την Επιτροπή. Ολοκλήρωσα, κυρία Πρόεδρε. Και ήταν σημαντικό να υποθούν αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά να τα λέμε σύντομα, λέει η Πρόεδρος, γιατί και άλλοι συναδελφοί έχουν ερωτήσεις. Ναι, αλλά εγώ είμαι συγκίτρια, λέει η κυρία Ριβασί. Λοιπόν, ε, καταρχήν να δώσω το λόγο στον Επίτροπο για να απαντήσει και μετά ε, θα απαντήσω και εγώ, θα τοποθετηθώ και εγώ ε, στα δικά μου τα θέματα. Ο Επίτροπος καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ την κυρία Βουλευτή για τα σχόλιά της, για τις συστάσεις της, ε, για όλα αυτά που είπε σε σχέση με την χρήση των κονδυλίων των φορολογουμένων όταν πρόκειται για ε, εξωτερικές δράσεις. Νομίζω ότι πρέπει να βελτιώσουμε την, ε, το πώς επικοινωνούμε τις εξωτερικές δράσεις, γιατί Όσον αφορά στη διαχείριση των προγραμμάτων μας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είναι εμφανής η δράσεις μας. Εγώ οποτεδήποτε ταξίδεψα στην Αφρική και οποτεδήποτε εφαρμόζονται προγράμματα ε, βλέπει κανείς πινακίδες ε, με το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί κανείς να μιλήσει με την κυβέρνηση ε, και να ξέρει ότι αυτό είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά όταν εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα κυρίως με διεθνείς οργανισμούς, τότε πράγματι δεν είμαστε τόσο εμφανείς Προσπάθησα να εξηγήσω στους συνομιλητές μας, στις κυβερνήσεις, ότι όταν ομιλούν για την υποστήριξη που έχουν από την Παγκόσμια Τράπεζα ή από τους φορείς των ΗΕ, τους λέω, τουλάχιστον το 40% αυτών των προγραμμάτων χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δηλαδή, ένα μεγάλο κομμάτι είναι δικά μας χρήματα. Αλλά αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το πούμε απευθεία στις ε, κυβερνήσεις. Κατά τα άλλα πρέπει να είμαστε περισσότερο εμφανείς, να φαινόμαστε, φαινόμαστε περισσότερο και να έχουμε πιο ουσιαστικό στρατηγικό διάλογο με τους ε, διεθνείς οργανισμούς. Τα έγγραφα ε, πολιετούς ε, συνεργασίας, τα έγγραφα που καθορίζουν αυτή την οικονομική συνεργασία, αυτά ε, θα πρέπει να περιλαμβάνουν κάποιες ρήτρε που να λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να φαίνεται να φαίνεται περισσότερο, να φαινόμαστε περισσότερο από όλους. Τώρα, όσον αφορά στην εξάλληψη της φτώχειας, Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι πράγματι ε, στο πώς ε, κάνουμε εμείς την οικονομική συνεργασία. Αν δείτε την Ευρωπαϊκή Συνένεση για τη συνεργασία και το περιεχόμενο και τη φύση των προγραμμάτων μας, η εξάλληψη της φτώχειας βρίσκεται στο κέντρο των προσπαθειών μας. Και έτσι θα συνεχίσει να είναι. Γιατί αυτή είναι η ευθύνη μας. Αυτή η ευθύνη απορρέει από τα, τους στόχους της χιλιετίας. Η εξάλληψη της φτώχειας βρίσκεται στην καρδιά αυτών των στόχων της χιλιετίας. Και νομίζω αυτό θα παραμείνει έτσι. Θα είναι απόλυτα ορατό ε, και στις δικές μας τις δεσμεύσεις. Συμφωνώ επίσης μαζί σας ότι δεν θα έλεγα ότι πρέπει να σταματήσουμε να μετράμε τα κονδύλια που εκταμιεύουμε για την αναπτυξιακή συνεργασία, αλλά θα έλεγα ότι οφείλουμε να βρούμε ε, έναν διαρθρωμένο, συστηματικό τρόπο για να μπορούμε να μετράμε το αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου Πράγματι ασχοληθήκαμε με τη μεθοδολογία, με το πλαίσιο, με τους στόχους, τους δείκτες που θα μας επιτρέψουν να παρουσιάσουμε σε όλους ε, τι ακριβώς επιτύχαμε με τη χρηματοδότηση, την αναπτυξιακή χρηματοδότηση σε εταιρικές, ε, σε χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Έχουμε σημειώσει πρόοδο στο να καθορίζουμε τα δεδομένα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στο να είμαστε πιο ορατοί, πιο εμφανείς ε, στα αποτελέσματα. Για τους μηχανισμούς ελέγχου και πάλι θέλω να σας πω ότι αυτοί αναφέρονται στους οικονομικούς μας κανόνες Υπάρχουν αρκετές φάσεις μηχανισμών ελέγχου στα προγράμματα μας ε, αναπτυξιακής συνεργασίας, Στα κεντρικά μας γραφεία, στην ΤΕΦΚΟ, έχουμε μία αντιπροσωπεία, έχουμε ε, το ελεγκτικό συνέδριο, στο κοινοβούλιο, αλλά πράγματι συμφωνώ ότι θα πρέπει να συνεργαζόμαστε περισσότερο και να συμπεριλαμβάνουμε και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Να μην είναι ναι, μόνο οι εταίροι μας κατά την εφαρμογή, αλλά εταίροι και στον έλεγχο, στην εποπτεία στο να καλούν σε λογοδοσία όλους όσοι συμμετέχουν στην ε, διαδικασία ανάπτυξης. Πάμε τώρα στα καταπιστευματικά ταμεία. Αν έχετε καλοσύνη μπορείτε να σταματήσετε γιατί μέχρι τώρα έχετε μιλήσει ήδη έξι λεπτά. Ε, πέντε λεπτά είχα προβλεφθεί για εσά και υπάρχουν και πολλοί άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να λάβουν το λόγο. Ε, κοιτάξτε για τα καταπιστευματικά ταμεία θέλω να σας πω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε ταχύτεροι και καλύτεροι χρησιμοποιώντας τα καταπιστευματικά ταμεία, ε, τις μεθόδους εφαρμογής. Τα καταπιστευματικά ταμεία ε, τα αιτήματα έρχονται από εδώ. Αυτό ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια όταν ε, είπαμε ότι δεν θα πρέπει να απευθυνόμαστε στους διεθνείς οργανισμούς, αλλά να χρησιμοποιούμε περισσότερα τα δικά μας, τα καταπιστευματικά ταμεία. Άρα δηλαδή ε, δεν θα πρέπει να ε, διωγγώσουμε όλη αυτή την κατάσταση σχετικά με τα καταπιστευματικά ταμεία, αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι τώρα βοηθούν στο να μας προσφέρουν τη δυνατότητα να ε, δημιουργήσουμε τη σωστή ισορροπία, το συσχετισμό με τη μετανάστευση και την ε, αναπτυξιακή μας ατζέντα. Αυτά θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον. Πολύ ωραία κύριε Επίτροπε. Λοιπόν, τώρα να προχωρήσω και εγώ με τις δικές μου τις ερωτήσεις. Καταρχήν, όσον αφορά στη συνεργασία με την Επιτροπή Αφρικανικής Ένωσης. Η Επιτροπή στο θέμα αυτό έχει εκφράσει μία επιφύλαξη και η Επιτροπή Αφρικανικής Ένωσης ε, συμμετέχει στην διαχείριση του εργαλείου African Peace για την Αφρικανική Ειρήνη. Ε, θα ήθελα να γνωρίζω πού ακριβώς ε, αναφέρεται η επιφύλαξη και τι ακριβώς πρέπει να γίνει έτσι ώστε να αρθεί η επιφύλαξη αυτή. Ερώτημα υπαριθμών 2 αφορά στη συνεργασία με τους αποκαλούμενους implementing partners, εταίροι κατά την εφαρμογή. Πώς μπορεί να βελτιωθεί η συνεργασία με το ελεγκτικό συνέδριο. Ε, πρέπει να σας πω ότι είμαι αρκετό καιρό στην Επιτροπή Ελέγχου Προεπλογισμών, παλαιότερα μέλος, μετά αντιπρόεδρος, αντιπρόεδρος τώρα πρόεδρος ε, και ε, τότε είχαμε πει ότι Δυστυχώ υπάρχει δυσκολία στην εργασία με την UNICEF και την DUEN και τώρα ισχύει πάλι το ίδιο. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω πώ μπορούμε να καταλήξουμε σε μια καλή μορφή συνεργασία. Ε, και επειδή και εμείς είμαστε βασικός χρηματοδότης των Ηνωμένων Εθνών, ε, θα πρέπει και τα Ηνωμένα Έθνη να δεχτούν ότι ε, και το ελεγκτικό συνέδριο και εμείς θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε κατά πόσον εκταμιεύονται σωστά τα κονδύλια. Να επαναλάβω και την ερώτηση της κυρίας Ριβάζη σχετικά με, τους, με τον εξαναγκασμό σε εργασία. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα χρηματοδοτούνται δεν είναι τέτοια φαινόμενα, φαινόμενα εξαναγκαστικής εργασίας. Θα ήθελα να έχω μια ξεκάθαρη απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν το κατάλαβα καλά, αλλά επειδή εσείς το είπατε με αφορά όμως και εμένα, το ξαναθίγω αυτό το θέμα. Κατόπιν θα ήθελα να έχω μία απάντηση για την μελέτη σχετικά με το υπολοιματικό ποσοστό σφάλματος. Η Κομισιόν αναφέρεται σε μία μελέτη του 2006. Πώς είναι δυνατόν σε αυτή τη μελέτη για το υπολοιματικό ποσοστό σφάλματος. Ε, είμαστε στο 18 και μου παρήσε ξαφνικά αυτή η μελέτη του 2006. Δηλαδή πριν από 12 χρόνια. Μήπως υπάρχει κάποια αιτιολογία ε, τι ακριβώς είναι αυτό το project όπου πρέπει να ε, ανατρέξουμε στο 2006. Κατόπιν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ε, υπέγραψε μία συμφωνία πλαίσιο με τα Ηνωμένα Έθνη και τώρα προσβλέπει στην αναβάθμιση του όρου reference, την αναφορά για τη συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Με συγχωρείτε, στην αναβάθμιση του όρου terms of reference, ε, μέσα αρμοδιοτήτων. Μήπως μπορείτε να μας εξηγήσετε λιγάκι τι ακριβώς εννοείτε με αυτό το θέμα σχετικά με τον ε, τομέα αρμοδιοτήτων. Η κυρία Ρίβαζη είπε επίσης ε, το πώς ακριβώς μπορούμε να μετρήσουμε την επιτυχία μας ποσοτικά. Η μέθοδος που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή να μετράτε ποσοτικά την επιτυχία. Ποια είναι αυτή η μέθοδος, ας πούμε, σε θέματα ε, φυγής από εμπόλεμες καταστάσεις, ε, σε θέματα εξάλληψης τόχιας. Δεν το έχω καταλάβει. Πώς ακριβώς το μετράτε αυτό ποσοτικά. Και θα ήμουν ευγνώμων αν μπορούσατε να απαντήσετε σε όλα αυτά προς την ΕΚΑ ε, και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω και εκεί κάποιες ερωτήσεις για την Global Europe παγκόσμια Ευρώπη. Εκεί δεν έχουμε συγκεκριμένα ποσοστά σφάλματος. Ποιο θα έπρεπε να είναι το δείγμα για να περάσουμε σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό σφάλματος. Αυτό είναι ένα ερώτημα προς την Επιτροπή και προς την ΕΚΑ και κατόπιν όσον αφορά στο ποσοστό σφάλματος 5,2 Βεβαίως γνωρίζω πολύ καλά ότι εργαζόμαστε σε δύσκολους τομείς. Όσον αφορά την ΕΚΑ που ανέφερα προηγουμένως, εννοούσα το ελεγκτικό συνέδριο. Με συγχωρείτε. Ε, θα ήθελα επίσης να πω ότι εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσοστά τα οποία πράγματι διαφοροποιούνται πάρα πολύ από αυτά που ανέφερε η Επιτροπή. Ως εκ τούτου, μία ερώτηση και προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποια μέτρα λοιπόν πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε αυτό το ποσοστό σφάρματος του 5,2 που είναι πάρα πολύ σημαντικό να μειωθεί το ποσοστό αυτό. Κατανοώ βέβαια την Επιτροπή που λέει ότι προέβησε διορθώσει, διορθώσεις. Ε, βλέποντας όμως ποια ποσά μπορούμε να ανακαλέσουμε, βλέπω ότι τα ποσά που μπορούν να κληθούν είναι πολύ περιορισμένα. Ως τούτου ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να δουλέψουμε λιγάκι στις ε, δομές. Και γι' αυτό θέλω να σας παρακαλέσω να μας πείτε από αυτό το 5,2% ε, κατά την άποψή σας πώς μπορούμε να κατέβουμε. Αυτά είχα να σας ρωτήσω και ευχαριστώ. Κύριος Επίτροπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Σε ό,τι αφορά την επιφύλαξη για το πρόγραμμα εφαρμογή της Αφρικανικής Ένωση. Ναι, η Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωση είναι σημαντικός ε, εκτελεστικό εταίρος. Αυτό ισχύει εδώ και πολλά χρόνια, κυρίως ε, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του μηχανισμού για την ειρήνη στην Αφρική. Και αυτό που μας ανησυχούσε συνεχώς ήταν το γεγονός ότι δεν ήμασταν σίγουροι ότι η Επιτροπή οι ικανότητε μάλλον της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωση, κυρίω σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, θα μπορούσαν να μας δώσουν ε, μια αξιόπιστη αποτίμηση σχετικά με τη χρησιμοποίηση της συνεισφοράς ε, για το μηχανισμό για την ειρηνή στην Αφρική. Έτσι λοιπόν, σε πολλές ε, συμφωνίες, σε έγγραφα, προσπαθήσαμε να έχουμε τη διαβεβαίωση ότι η Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης θα μπορούσε να εφαρμόσει τα προγράμματα του Μηχανισμού για την Ειρήνη στην Αφρική στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο των προτύπων για τον έλεγχο και της εφαρμογής. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να επιταχύνουμε την αξιολόγηση των έξι πυλώνων της Επιτροπής Αφρικανικής Ένωσης. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία είναι υπό εξέλιξη. Μπορεί να καταλήξει και είμαστε θετικοί ότι σε ένα μήνα θα μπορούσαμε να έχουμε μια οριστική επιβεβαίωση ότι η Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης έχει βελτιώσει τις ικανότητές της, ε, κυρίως ε, για να διεξάγει τις διαδικασίες ε, δημοσίων συμβάσεων βάσει προτύπων. Αν επιβεβαιωθεί αυτό από την αξιολόγηση των πυλώνων, θα αποσύρουμε την επιφύλαξη σε σχέση με την Επιτροπή αυτή. Τώρα, οι εταίροι της ε, εκτέλεσης ε, των προγραμμάτων ε, και ιδίω οι διεθνείς οργανισμοί είναι οι εταίροι μας. Σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουμε τα ίδια προβλήματα που έχουμε με την Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης, παραδείγματος χάρη. Υπάρχει αξιολόγηση πυλώνων για όλους, υπάρχουν οι συμφωνίες πλαισίου, και τα μνημόνια συνεννόησης, με την Παγκοσμία Τράπεζα, με τους ε, φορείς της υπηρεσίας του ΙΕ κτλ. Όμως εξακολουθεί να υπάρχει ένα πρόβλημα, κυρίως σε ό,τι αφορά την ε, παροχή των απαραίτητων εγγράφων, ιδίως για τις διαδικασίες ελέγχου. Φέτος, είχαμε έναν ε, σημαντικό παράγοντα. Αυτό ήταν μάλλον ένα σημαντικός παράγοντας και αυτό αύξησε το επίπεδο σφάλματος και φτάσαμε σε αυτό το απαράδεκτο ποσοστό σφάλματος του 5,2%. Όμως ε, δεν μιλάμε για μια ξαφνική αλλαγή της πολιτικής ή της πολιτικής βούλησης των διεθνών οργανισμών να παράσχουν τα έγγραφα. Ουσιαστικά αποτελεί ένα μείγμα αιτιών. Δηλαδή ότι μπορεί να είχαμε μικρότερη περίοδο που δόθηκε στους διεθνείς οργανισμούς να δώσουν τα έγγραφα αυτά. Αλλά φυσικά όλα αυτά δεν αιτιολογούν τη συμπεριφορά και την βραδύτητα με την οποία παρέχουν τα έγγραφα οι διεθνείς οργανισμοί. Έτσι λοιπόν στις υπηρεσίες ΤΕΦΚΟ αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε πλήρως τις συστάσεις του Λεκτικού Συνεδρίου και να εργαστούμε πιο άμεσα με τους διεθνείς οργανισμούς, να τους παρέχουμε και ένα είδος τεχνικής βοήθειας, προκειμένου να τους αναγκάσουμε να μας παρέχουν τα απαραίτητα έγγραφα εγκαίρως. να πληρούν δηλαδή τις υποχρεώσεις τους ε, που αναφέρονται σαφέστατα στις συμφωνίες. Έχουμε λοιπόν αυτό το κοινό εγχείρημα πολύ περισσότερο τώρα από ό,τι στο παρελθόν. Και επίσης προωθούμε τον διαρθρωτικό διάλογο και τον ετήσιο διάλογο μαζί τους προκειμένου το θέμα αυτό να μπει στην κορφή του κοινού μας θεματολογίου. Κύριε Επίτροπε, σε πέντε λεπτά Σα είχα ζητήσει να απαντήσετε, δηλαδή μιλάτε ήδη πέντε λεπτά και δεν έχετε απαντήσει ακόμα. Θα ήθελα να απαντήσετε γραπτό και κυρίω ό,τι αφορά την καταναγκαστική εργασία. Ναι, θα δώσουμε και γραπτέ απαντήσει ό,τι αφορά του όρου αναφορά για του διεθνεί οργανισμού. Σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία και το πώς υλοποιείται το πλαίσιο αποτελεσμάτων, θα δώσουμε τις απαντήσεις ε, γραπτώς. Και... Κυρία θα θέλει πρώτα το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, σκιώδης και για τα δύο θέματα και θα μιλήσω και για τα δύο. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ για το έργο σας τα τελευταία πέντε χρόνια και ευχαριστούμε για τις απαντήσεις που μας δίνετε. Επίσης ευχαριστώ και το ελεγκτικό συνέδριο και κυρίως ε, την παρουσίαση για τις ε, εκθέσεις. Για την απαλλαγή της Επιτροπής πρώτα απ' όλα. Ζητώ συγγνώμη γιατί καταλαβαίνω ότι υπήρξαν κάποια θέματα ε, και οι ερωτήσεις μας ε, κάποιες δεν έφτασαν στο γραφείο σας. Κάποιες είναι λεπτομερείς, οπότε σας παρακαλούμε να τις ξαναστείλουμε και να έχουμε γραπτά τις απαντήσεις. Μία από αυτές τις ερωτήσεις θα θέσω τώρα. Και γραπτά μπορείτε να τη συμπληρώσετε την απάντησή σας. Λοιπόν, σύμφωνα με το σχέδιο εργασίας για το 2019 όσον αφορά τους διεθνείς οργανισμούς που συζητάμε, ο ορισμός διεθνείς διεθνής οργανισμός περιλαμβάνει και άλλες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που ε, θεωρούνται συναφείς με τους διεθνείς οργανισμούς. Μπορείτε σας παρακαλώ να μας πείτε ποια ακριβώς είναι τα κριτήρια ε, βάσει των οποίων πήρε αυτή την απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πότε την πήρε αυτή την απόφαση. Και θέλουμε επίση περισσότερε διευκρινήσει για το πόσε αποφάσει πήρε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, σα είπα και γραπτά θα σα στείλουμε τι ερωτήσει μα, γιατί θέλουμε λεπτομέρειες. Αυτή είναι η ερώτησή μου για την απαλλαγή όσον αφορά την Επιτροπή και τώρα περνάω στο EDF, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Οι γραπτές σας απαντήσεις είναι αρκετά λεπτομερείς. Ε, κάποια σχόλια έχω όσον αφορά την ερώτηση αριθμός 1. Πρώτα απ' όλα, στο 1α λέτε ότι διάφορες κυρώσεις θα μπορούσαν να επιβληθούν εφόσον μια οργάνωση εταίρος δεν δίνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε κατά πόσο τέτοιες κυρώσεις έχουν ποτέ εφαρμοστεί και πότε ήταν τελευταία φορά που εφαρμόστηκαν τέτοιες κυρώσεις. <clears throat> Επιβλήθηκαν τέτοιες κυρώσεις. Έπειτα στο ένα β για την ερώτηση α πάντα. Εξηγείται ε, το ποσοστό σφάλματος και λέτε ότι πολλές φορές οφείλεται σε έλλειψη δικαιολογητικών από διεθνείς οργανισμούς και έπειτα φταίει και το ότι δεν υπάρχει πάντα αρκετός χρόνος ε, σε σχέση και με τον έλεγχο από το Ελληνικό Συνέδριο, το οποίο και θέλω να ρωτήσω, θα μπορούσατε να δώσετε ε, μεγαλύτερα περιθώρια ώστε να μην έχουμε τέτοια ε, σφάλματα που οφείλονται στην έλλειψη χρόνου. Κατά τα άλλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την διαφάνεια. Εκεί που στην απάντηση στην ερώτηση 1 λέτε ότι υπάρχει και ιδιαίτερα ε, υψηλό φόρτο εργασίας και όχι αρκετό προσωπικό. Συχνά δεν έχουμε τέτοια απάντηση από άλλα ε, όργανα, οπότε ευχαριστούμε για τις απαντήσεις σας αυτές, τις τόσο ανοιχτές και ελεύθερες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε πίτροπε για τα σχόλιά σας και τις απαντήσεις σας. Εγώ θέλω να θίξω διάφορα ζητήματα. Πρώτον, το θέμα της έλλειψης συνεργασίας ε, με την Αφρικανική Ένωση. Εσείς στην αρχή αναφερθήκατε στην προθεσμία που έχει στη διάθεσή του κάθε διεθνής οργανισμός και φαίνεται ότι έχουν πάρα πολλή δουλειά να κάνουν μέσα σε αυτά τα περιθώρια τα χρονικά για να ανταποκριθούν σε αυτά που ζητάτε. Έπειτα η Αφρικανική Ένωση προφανώς έχει λιγότερο προσωπικό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις προθεσμίες με τόσο περιορισμένους πόρους. Οπότε είπατε ότι θα μπορούσε να υπάρξει βελτίωση εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο πυλώνας στο τέλος. Αν όμως δεν υπάρξει τέτοια βελτίωση, τι σχέδιο έχετε η Αφρική Ένωση τι θα κάνει με την αξιολόγηση του πυλώνα. Και η τελευταία μου ερώτηση έχει να κάνει με την απάντησή σας στις γραπτές ερωτήσεις στη σελίδα 11. Υπάρχει η ερώτηση για το κίνδυνο να υπάρξει εμπορικός πόλεμος με την Κίνα. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην αναπτυξιακή βοήθεια είναι σίγουρα πολύ διαφορετική από ό,τι αυτή της Κίνας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι δημοκρατική οργάνωση και έχει μια δημοκρατική προσέγγιση, ενώ αντίθετα η Κίνα έχει μια περισσότερο αυταρχική στάση. Οπότε στην πράξη εσείς Βλέπετε η δικιά μας η αντιμετώπιση η ήπια αυτή η προσέγγιση να βοηθάει, δεδομένου ότι η προσέγγιση όπως είπαμε Κίνας και Ευρώπης, που δεν είναι συμπληρωματικές, είναι μάλλον ανταγωνιστικές μεταξύ τους, μια που εμείς ζητάμε να τηρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, αξιολόγηση πυλώνα κλπ. Η Κίνα δεν ζητάει τέτοια αξιολόγηση πυλώνων. Δίνει χρηματοδότηση Πώς τοποθετείτε λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει αποτελέσματα καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ, Βιόλα Φων ε, Κράμα. Ευχαριστώ πολύ, ε, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, επειδή δεν έχουμε ε, αρκετό χρόνο, σε 10 λεπτά πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μου απαντήσετε γραπτά σε αυτά που θα σας ρωτήσω ή δυνατόν. Και η ερώτησή μου είναι η εξή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις αρχές της Λιβύης και μία σειρά διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στη Λιβύη. Υπάρχουν αρκετές εκθέσεις σχετικά όμως με ε, καταχρήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από τις τοπικές αρχές στη Λιβύη. Ε, σε γραπτή απάντηση αναφέρεται ότι η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει εσωτερικό έλεγχο, αλλά για λόγους ασφαλείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εξωτερικό έλεγχο. Και η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξή. Οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αναφέρουν στα συστήματα εσωτερικών ελέγχων ε, κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Επιτροπή μπόρεσε να παρακολουθήσει τα προγράμματα που αναφέρονται εσωτερικά ή από άλλους οργανισμούς όπως είναι ΜΚΟ και άλλα μέσα και επιπλέον στην απτή απάντησή λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να αυξήσει αυτές τις προσπάθειες προσπαθώντας να επαληθεύσει όλα όσα έχουν επιτευχθεί στη Λιβύη. Τέλος της παράθεσης. Μήπως μπορείτε λιγάκι να διευκρινίσετε τι είδους προσπάθειες ε, θα λάβουν χώρα και πώς μπορεί να αποφευθεί μια κατάσταση όπου οι αρχές της Λιβύης που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε πολλές περιπτώσεις ε, πράγματι Ισχύει αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω στους συναδέλφους ότι στις ε, γραπτές ε, ερωτήσεις ε, με συγχωρείτε, μια παρατήρηση εκτό μικροφώνου. Συνεχίζει η πρόεδρο. Βιόλα, αν έχετε καλοσύνη, αφήστε με να ολοκληρώσω. Διακόπτει η μιλήτρια, αλλά δυστυχώ εκτό μικροφώνου. Ε, εγώ λέω να δώσουμε το λόγο σε όλους και κατόπιν να τεθούν και ερωτήσεις προς τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ. Γιατί εδώ δεν έχουμε χρόνο. Αυτή τη δυνατότητα ήθελα να προσφέρω σε όλους τους ε, ε, συμμετέχοντες. Παρακαλώ και μετά ο κύριος Μίμικα. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάλφοι, σήμερα δεν έχουμε χρόνο. Γι' αυτό εγώ ε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και θα υποβάλω τις ε, ερωτήσεις μου. Είδα λιγάκι τις ε, εκθέσεις. Ε, πάω πίσω, πήγα πίσω πέντε χρόνια πίσω. Και νομίζω ότι προσπαθείτε πράγματι αλλά παρόλα αυτά ε, υπάρχει ένα υψηλός, υπάρχει υψηλός κίνδυνος σφάλματος. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας ερωτήσω, θέλετε να εισάγετε ένα σύστημα αξιολόγησης εξάντε όπου εντοπίζονται τα προγράμματα τα οποία συνοδεύονται με υψηλό κίνδυνο πριν ε, ε, επενδυθούν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ σε σχέση με τη δυνατότητα να εξομοιώσουμε κάποιες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις με διεθνείς οργανισμούς. Τα κριτήρια μεθοδολογίας τίθεται από τους νομοθέτες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και οι σχετικούς δημοσιονομικούς κανόνες. Και επίσης παρέχονται γραπτός στις απαντήσεις μας στην Επιτροπή. Όμως υπάρχει μόνο μία μη κερδοσκοπική οργάνωση με την οποία, μάλλον την οποία εξομοίησε. Η Κομισιόν πρόκειται για το Παγκόσμιο Ταμείο την κατεπολέμηση της ελληνοσίας ε, του AIDS και της φυματίωσης σε σχέση με το σέβεται τα κριτήρια των κανονισμών. Τώρα, για τη μην παροχή των δικαιολογητικών. Προτιμάμε να συνεργαζόμαστε με τους διεθνείς οργανισμούς, με τους εταίρους μας, με τον τρόπο που προσπάθησα να σας εξηγήσω. Δηλαδή να τους καταστήσουμε πιο ταχείς και πιο έτοιμους να μας δίνουν εγκαίρους τα δικαιολογητικά. Όταν όμως είναι προφανές ότι μια τέτοια προσέγγιση δεν ωφελεί, Λαμβάνουμε όλα τα άλλα μέτρα που έχουμε στους χρηματοοικονομικούς κανονισμούς. Με το σχάρι με το φόρουμ για τον ειρηνικό. Όπου σταματήσαμε τη χρηματοδότηση ορισμένων προγραμμάτων επειδή δεν μας είχαν δώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τώρα για την Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης. Ναι, συνεργαζόμαστε μαζί της ε, και ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια θετική αξιολόγηση. Αλλά αν όχι, και ακόμη και πριν το θετικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης πυλώνων, σε ορισμένες περιπτώσεις αλλάξαμε τον εταίρο μας. Παραδείγματο χάρη στο να υποστηρίξουμε τις κοινέ δυνάμεις στο ΣΑΧΕΛ, ε, θα εφαρμοζόταν αυτό το project από την Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης αλλάξαμε τον εταίρο μας ε, και ήρθαμε σε επαφή με την Expertise France. Γιατί αυτός ο οργανισμός μπορούσε να μας δώσει περισσότερες εγγύησεις ότι θα εφαρμοστούν αυτά τα προγράμματα. Αυτό θα ισχύει και για το μέλλον. Ελπίζουμε η Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης να τα πάει καλά στην αξιολόγηση πυλώνων. Για τις σχέσεις με την Κίνα. Ναι, Πολύ διαφορετικά υλοποιούμε την αναπτυξιακή συνεργασία, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε τη δική μας οδό. Η δική μας αναπτυξιακή συνεργασία δεν καθορίζεται από το τι κάνουν ή δεν κάνουν οι άλλοι. Ε, το δική μας αλληλεγγύη καθαρίζεται από το γεγονός ότι είμαστε ο μεγαλύτερος πάροχος ε, αναπτυξιακής βοήθειας. Με την Κίνα προσπαθούμε να μειώσουμε το χάσμα μεταξύ ανταγωνισμού και συμπληρωματικότητας των αναπτυξιακών προγραμμάτων μας. Είναι μακρά η διαδικασία αυτή. Δεν θα ήθελα να ισχυριστώ τώρα ότι είμαστε σωστοί εδώ και λαμβάνουμε περισσότερη υποστήριξη από την Κίνα σε αυτό. Κύριε Επίτροπε, συγγνώμη, πρέπει να σας ε, διακόψω. Ε, τις ε, πρέπει, τις ερωτήσεις πρέπει να τις απαντήσετε γραπτά. Ε, λυπάμαι πάρα πολύ. Ε, ζητώ συγγνώμη, αλλά απευθύνομαι και στα μέλη των Σε δύο λεπτά πρέπει να ε, γίνει η ψηφοφορία και οι συνάδελφοι πρέπει να φύγουν. Σε δύο λεπτά αρχίζει η ψηφοφορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.